Μπορείτε να καθίσετε όλοι, ιδίως ο Μάρκους Πίπερ. Γιατί έχουμε πλήρη ημερησία διατάξη. Καλό απόγευμα σε όλους. Ε, η συνεδρίασή μας μεταδίδεται και στο διαδίκτυο, όπως ξέρετε, και σε σχέση με την ημερησία διάταξη, δεν είναι ικανοποιημένη με την ημερησία διάταξη, θέλω να την αλλάξουμε. Θα σας προτείνω κάποιες αλλαγές λοιπόν. Η πρώτη αλλαγή σε σχέση με την έκθεση του κυρίου Λούχαν για την εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως απαράγραπτη προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα. Συμφωνήθηκε μεταξύ των συντονιστών να αναβληθεί η ψηφοφορία για την έκθεση αυτή μέχρι την επόμενη συνεδρίασή μας λόγω μιας πλημμυρόδου ροής τροπολογιών που μας εμποδίσει να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Προτείνεται επίσης από τους συντενιστές να θέσουμε στη μέση διάταξη το σημείο 13α, δηλαδή ανταλλαγή απόψεων για την ε, γνωμοδότηση μας προς την Οικονομική Επιτροπή σε σχέση με ένα κανονισμό για την κρατική για την κρατικές βοήθειες για το κλείσιμο των μη ανταγωνιστικών ορυχείων και η άλλη αλλαγή αφορά την, ε, την έκθεση του κύριου Μποστινάρου που είναι γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σε σχέση με τη στρατηγική της Μαύρης Θάλασσας. Δεν υπάρχει καμία βιασύνη. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό σε μία από τις μεταγενέστερες συνεδριάσεις μας. Αν συμφωνείτε λοιπόν και αν δεν υπάρχει καμία άλλη αίτηση για αλλαγές, αμέσως κύριε Πίπερ, μπορούμε να δεχτούμε την τροποποιημένη ε, η Ο Μάρκους έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Θα ήθελα να ζητήσω κάτι για τις συνεδρίες των συντονιστών απόψε το βράδυ. Πρόκειται για την έκθεση ΑΕΠ και επέχεινα και πιστεύω ότι η αρχική αρμοδιότητα για την περιφερειακή ανάπτυξη, την ευμάρεια σε ε, περιφερειακό επίπεδο και για την καταμέτρηση της ε, ανάπτυξης και της ευμάρειας είναι αρμοδιότητα της δικής μας Επιτροπής και όχι της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο έχει γίνει επίτηδες στη συγκεκριμένη περίπτωση, στοχευμένα, γιατί οι εισηγητέ είναι όλοι πράσινοι σε αυτήν την περίπτωση. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό όπως αυτή η έκθεση η οποία αφορά τις κεντρικές μας, τις κομβικές μας αρμοδιότητες, το θέμα του ΑΕΠ ως δίκτυ, να περάσει σε κάποια άλλη επιτροπή. Θα ήθελα να συζητήσουμε λοιπόν απόψε το βράδυ, μήπως θα ήταν δυνατό αυτή η έκθεση να έλθει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Θα είμαστε εμείς αρμόδια επί της ουσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πράγματι αυτό το θέμα βρίσκεται στην ημέρησια διαταξή μας αύριο. Για αύριο, αν καταλήξουν λοιπόν οι συντονιστές σε κάποια απόφαση που απαιτεί και τροποποίηση της ημερησίας διάταξης, θα μπορέσουμε να κάνουμε εκεί πέρα και μια αλλαγή ακόμα. Και για τη συνεδρίαση των συντονιστών θέλω να σας υπενθυμίσω ποιο είναι το ιστορικό για το θέμα αυτό, γιατί υπήρξε μακρά συζήτηση τον Οκτώβριο του 2009 και η συζήτηση αυτή κατέληξε στην τρέχουσα απόφαση. Μπορούμε να επανέλθουμε στο θέμα αυτό στη συνεδρίαση των συντονιστών. Εάν δεν υπάρξει λοιπόν κάτι άλλο το οποίο θέλετε να εγγύρετε θεωρώ ότι έχει εγκριθεί η ημερήσια διάταξη με την δυνατότητα μετά από τα σχόλια του Μάρκους Πίπερ να υπάρξει κάποια αλλαγή για το θέμα αυτό του ΑΕΠ και θέλω να σας πεθυμίσω ότι τη ψηφίσουμε αύριο στις 9 ακριβώς. Σας παρακαλώ να φέρετε τις κάρτες ψηφοφορίας για αύριο. Και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξης που είναι η έγκριση του σχεδίου χρονοδιαγράμματος για τις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής κατά το έτος 2011. Έχετε στο φακελό σας το χρονοδιάγραμμα αυτό. το χρονοδιάγραμμα του Κοινοβουλίου καταρχήν που προετοιμάστηκε από τις υπηρεσίες του και καταρχήν λαμβάνει υπόψη τη διαθεσιμότητα δωματίων αιθουσών συνεδριάσεων και επίσης διερμηνέων, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη γλωσσική διάσταση της Επιτροπής μας. Έχετε λοιπόν αυτό το χρονοδιάγραμμα. 11 τακτικές συνεδριάσεις έχουμε και έχουμε φυσικά και το δικαίωμα να κάνουμε και έκτακτες συνεδριάσεις οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί στο τρέχον αυτό χρονοδιάγραμμα και μπορείτε να δείτε ότι οι περισσότερες συνεδριάσεις μας είναι στην αρχή της εβδομάδας, Δευτέρα Τρίτη ή Δευτέρα Τετάρτη. Μέχρι τώρα οι συνεδριάσεις μας ήταν δύο μισές μέρες. Αλλά μπορεί να υπάρξουν και αλλαγές σε αυτό, να έχουμε συνεδριάσεις μισής μέρας και άλλες συνεδριάσεις που κάνουν μια μισή μέρα, τρεις μισές μέρες. Κατά μέσον όρο οι συνεδριάσεις μας όμως θα διαρκούν δύο μισές μέρες. Αν μπορείτε λοιπόν να εγκρίνετε και αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης, θα περάσουμε στο επόμενο, η ανακοινώσει της Προέδρου. Και εδώ θα ήθελα να σας ε, αναφέρω ποιες ήταν οι αποφάσεις των συντονιστών στη συνεδρίασή μας της 6ης Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο. Αποφάσισαν τότε οι συντονιστές να προτείνουν τις εξής γνωμοδοτήσεις οι οποίες θα πρέπει να συνταχθούν από τα μέλη των, της Επιτροπής μας. Καταρχήν, για την ε, αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα που είναι αρμόδια η Επιτροπή Βιομηχανίας. Η γνωμοδότηση αυτή πάει στην κυρία Κολάσκα Πομπίνσκα στην ομάδα του ΕΛ. Η δεύτερη έκθεση πρωτοβου... γνωμοδότηση μάλλον σε μια έκθεση πρωτοβουλίας είναι για τη βιομηχανική πολιτική σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, πάλι της Επιτροπής Βιομηχανίας ε, Έκθεση Πρωτοβουλίας. Οι Σοσιαλιστέ και οι δημοκράτες παίρνουν την έκθεση αυτή, ο Φραντσέσκο Ντεαντζέλη συγκεκριμένα, και επίσης με την γραπτή διαδικασία αποφάσισαν οι συντονιστές να προτείνουν δύο γνωμοδοτήσεις οι οποίες θα πρέπει να συνταχθούν από την Επιτροπή μας, καταρχήν για τις κρατικές επιδοτήσεις για την ε, για το κλείσιμο αντιοικονομικών ή μάλλον μη ανταγωνιστικών ανθρακοριχείων. Ο Γιάνν Μπριτζίνια είναι εδώ ο συντάκτης νομοδότησης και η Επιτροπή επί Οικονομική και Νομισματική και η δεύτερη περίπτωση αφορά την απόφαση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Έτος για την ενεργό Η Επιτροπή Απασχόλησης είναι η αρμόδια επί της και η γνωμοδότηση ε, θα πάει στο ΕΛΚ, αλλά δεν έχουμε ακόμα κάποιο όνομα συγκεκριμένο για αυτή την έκθεση. Αν δεν υπάρχουν σχόλια λοιπόν, παίρναμε στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης η ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Γιάννους Λεβαντόσκι, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και την χρηματοοικονομική σχεδίαση, τη δημοσιονομική μάλλον σχεδίαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 4.30 να ανταλλάξουμε απόψεις. Πιστεύω ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως αυτό το χρόνο και επομένως θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Επίτροπο όσο χρόνο θέλετε, άπλετο χρόνο έχετε για να, εξε... για να εξηγήσετε όλα τα θέματα τα οποία συνάπτονται με τα ζητήματα του προπολογισμού και θα σα ακούσουμε αδειμόνως και ασμένως. Και φυσικά θα ακολουθήσουν ερωτήσεις καθώς και απαντήσεις. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ, Ντανούτα, για την πρόσκληση και για την εξουσία που μου έδωσες. Είπες ότι ό,τι πω είναι καλό. Ευχάριστο να το λες αυτό. Δεν θα τιμήσω την Ντανούτα Χόμπνερ μιλώντας πολωνικά, να... και θα υποκληθώ στην δεσπόσα θέση των Αγγλικών. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και, και την αλληλουχία των γεγονότων, Μπαίνουμε σε καυτή εποχή όσον αφορά τον προϋπολογισμό στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και αυτό που έχουμε τώρα μπροστά μας, η... θα αναβληθεί η δημοσιονομική αναθεώρηση για τον Οκτώβριο, διότι θέλουμε να συναγάγουμε μαθήματα από την κρίση όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Τέλος Σεπτεμβρίου, 29 Σεπτεμβρίου, τις επόμενες μέρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Κάποιες προτάσεις αφορούν πολιτική συνοχής και τον προϋπολογισμό που θα πρέπει να είναι εργαλείο για κυρώσεις και όχι απλώς για εγγύσεις για δανειοδότηση. Αλλά αυτό ζητά αναθεώρηση δημοσιονομική που καθυστέρησε. Ήταν απόφαση με επίγνωση του Συμβουλίου που ενεκρίθη από, την, ε, από το Κοινοβούλιο και ανατέθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται να ενδιαφέρεται για αυτή την αναθεώρηση. Τα άλλα θεσμικά όργανα και εθνικέ αντιπροσωπείε ήδη κοιτάνε τι επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικές και τι θα γίνει μετά το 2013. Αυτό που θα είναι κάπως επίμαχο, όπως είδαμε και τον Αύγουστο, μέσω μια αθώα συνεντεύξεω είναι και το εξή. Δεν θέλουμε μόνο να εξετάσουμε τις δαπάνες, αλλά όπως είχε δοθεί και στην εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να δούμε και τι γίνεται με, το, τα έσοδα. Τι θα παρουσιάσουμε στο παράρτημα τη αναθεωρήσεω, Αυτό είναι ο στόχο, μου. Απαρίθμηση των ιδίων πόρων που θα μπορούσαν να μειώσουν τις εθνικές συνεισφορές που εισραίουν άμεσα στον προπολογισμό. Ξέρω ότι δεν είναι καθόλου δημοφιλές ζήτημα ή δύσκολο, αλλά είναι στην εντόλη ότι θα πρέπει να παρουσιάσουμε ουδέτερη έκθεση για τους ιδίους πόρους και όχι μόνο για τις δαπάνες, τις ίδιες δαπάνες. Μετά πάμε στο στατικικό έγγραφο περί συνοχής, που έχει κατεύθυνση προς το μέλλον, πάρα πολύ σημαντικό έγγραφο, αφορά τη δομή της πολιτικής σύνοχης μετά το 2013. Το ίδιο αφορά και την κοινή αγροτική πολιτική. Φέτος θα συζητηθεί, θα παρουσιαστεί. Γίνονται ήδη προετοιμασίες για πολιτές πλαίσιο. Είμαστε υποχρεωμένοι, υπέχουμε νομική υποχρέωση να παρουσιάσουμε το πρώτο νομοθετικό πακέτο για το επόμενο πολιτές πλαίσιο μέχρι το τέλος Ιουνίου 2011. Προσπαθούμε να πετύχουμε τη σωστή, το σωστό χρονικό συντονισμό γιατί αναμένονται και ανακοίνωση για τα στοιχεία μετά το 2013. Για να τα κάνουμε αυτά από κοινού σε ένα νομοθετικό πακέτο είναι μια λύση. Θέλουμε να δούμε αν θα υπάρξει και άλλο συντονισμός. Ε, εγώ υποθέτω ότι το 2011 θα πρέπει να αφορά επίσης και τη λιτότητα στα κράτη-μέλη, μεγαλύτερη λιτότητα, διότι το πολιτικό πρόγραμμα υποχρεώνει του Υπουργού Οικονομικών να προβλέπουν μεγαλύτερη λιτότητα για τους προπολογισμού το 2012, κάτι που συζητηθεί το 2011. Και όχι τώρα, βέβαια, να μην συζητηθεί τώρα. Υπέχουμε όμως νομική υποχρέωση εμείς. Πολιτές πλαίσιο. Θα ενταχθεί σε γενική ανακοίνωση, είτε το τέλος Ιουνίου ή λίγο νωρίτερα. πριν στείλουμε το πρώτο νομοθετικό πακέτο. Όλα εξαρτώνται από το κλίμα που θα επικρατεί, το πολιτικό. Θέλουμε να υπάρχει σωστή αλληλουχία γεγονότων, χωρίς απογοητεύσεις. Θέλουμε να βελτιωθεί ο Ευρωπαϊκός Υπολογισμός στο μέλλον. Αυτός είναι ο στόχος. Το τελικό νομοθετικό πακέτο θα πρέπει να υποβληθεί το 2011. Άρα πρέπει όλα να ξεκαθαριστούν μέσω των προτάσεων Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 2011, να ξεκινήσουμε τα διαπραγματεύσει. Ελπίζουμε επί Δανέζικη Προεδρία. Ε, και έχουμε και τι γαλλικέ προεδρικέ εκλογέ το 2012. Είναι σημαντικά πολιτικά γεγονότα και πάντα εκεί δημιουργούνται ζητήματα οικονομικά. Άρα οι Δανείοι θα έχουν ένα μήνα για να πετύχουν συμφωνία. θα μπορεί να κληρωθούν συζητήσεις με το Κοινοβούλιο που θα έχει αυξημένες βέβαια εξουσίες μέσω της συνθήκης Λισαβόνας. Και ελπίζουμε μην έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Έχουμε μάθει κάποια μαθήματα από την περίοδο 2004-2006. Δηλαδή ότι αν καθυστερούμε πολύ, οι αρχές των επομένων δημοσιονομικών προπτικών δεν εφαρμόζονται εγκαίρως. Το είδαμε και το 2007-2008. Άρα έχουμε πίεση χρονική. Τι θέλω να σας πω. Θέλουμε να δούμε ποια είναι η βούλη των θεσμικών οργάνων, αν έχουν καλή διάθεση. Στη διαδικασία του 2011, για τον προπολογισμό 2011. Επίκειται μετά την ανάγνωσή σας συνδιαλλαγή, τον Οκτώβριο συνδιαλλαγή μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο μεσάζων ούτως υπήρ μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Πρόκειται περί πρωτοτύπου και διαδικασία μοναδική ανάγνωση Πρέπει να δούμε ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί όσον αφορά τα θεσμικά όργανα. Όσον αφορά τη συνοχή, Είμαστε στην Ευρώπη μετά την κρίση. Αυτό έχει άμεση συνέπειση κρίση στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Πέρα από το μέσο για τον ισολογισμό, 50 δις έχουν διατεθεί εκεί. Ο ευρωπαϊκό υπολογισμό είναι και εγγύηση για ενδεχόμενα δάνεια στα πλαίσια του μηχανισμού σταθεροποίηση μέχρι 60 δισεκατομμύρια ευρώ για τι χώρε Ευρωζώνη. Ευέλικτη ερμηνεία τη συνθήκη τη Αβώνα είναι αυτή. Αλλά έχουμε συμμετοχή του ευρωπαϊκού προπολογισμού στο μηχανισμό σταθερότητα. Ποιο είναι το επόμενο. Ο ευρωπαϊκό προπολογισμό σαν ένα εργαλείο, εργαλειοθήκη για κυρώσει. Πολύ σημαντικό αυτό. Στόχο μα ποιο είναι οι κυρώσεις να μην συγκεντρώνονται στην πολιτική συνοχή και μόνο και τις μεταφορές να αφορά το θέμα, όχι μόνο τη συνοχή. Αλλιώς είναι θεωρητική η ποινή για χώρες που δεν χρησιμοποιούν τη συνοχή και που παραβιάζουν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Θα υπάρχει διασύνδεση μεταξύ σταθεροποίησης και πειθαρχία της Ευρώπης μετά την κρίση. Και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ευρωπαϊκός προπολογισμός για όλα αυτά. Εγώ δεν είμαι υπέρ αξιολογήσεως του μέλλοντος συναρτήσει λιτότητας. Οι Εθνικοί Υπουργοί Οικονομικών θέλουν μια παγιοποιηση συνοποίηση για να βελτιωθεί η εξοπιστία των χρηματοστικών αγορών. Εμείς θέλουμε να δώσουμε αποτελέσματα στους, ε, στο λαό, στους μαθητές, του Εράσμου, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε δικαιούχους οι οποίοι θα μπορούν να προωθήσουν το πνεύμα που καταπολεμά την κρίση. Μιλάμε για επενδύσεις. Αυτή είναι η φύση των ε, διαθετικών ταμείων. Ξέρετε πολύ καλά ότι η συνοχή είναι κάτι που σατευόμενο συνθήκη της αγώνας. Αφορά όχι μόνο οικονομική, κοινωνική, αλλά και εδαφική διάσταση. Θα είναι πρωταρχικό μέσο για να προωθεί την εδαφική διάσταση και να προωθεί πολιτικές. Όσον αφορά το μέλλον, είμαι σε επαφή με τον Ιωάννης Χάν, επίτροπο υπεύθυνο για το θέμα. Θα είμαι σε επαφή εγώ με την Επιτροπή Ρέτζη. Στις 13 Ιουλίου ετοιμάσατε ένα έγγραφο που εκφράζει τη θέση σας. Εγώ νομίζω ότι δεν και οι θέσεις μας όσον αφορά το όραμα ποια θα είναι η πολιτική συνοχή μετά το 2013. θα πρέπει να μιλάμε για ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική και όχι για α, δωρεά ποσών στους στοχούς συγγενείς της Ανατολής. Πρέπει να δούμε ποιες δυνατότητες δημιουργούνται και πιο πολύ να δούμε δυνατότητες από φραγμούς. Πρέπει σε πολλαπλά επίπεδα να κινηθούμε. 70% από πάνω 400 λειτουργικά προγράμματα αποφασίζονται και εφαρμόζονται περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σοφό αυτό. Λαμβάνουμε υπόψη τις περιφερειακών, των περιφερειακών αρχών με την ευρωπαϊκή δομή. Σε πολιτές πλαίσιο θα κινηθούμε. Πέντε χρόνια το συζητάμε. Εφτά χρόνια. Όπως τώρα. Ή δύο επί πέντε με διάμεση αναθεώρηση. Θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη περιφερειακή ε, πολιτική συνοχής. Το κοινωνικό ταμείο να είναι ορατό. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ένα τμήμα κοινωνικής οικονομικής συνοχής στο τοπικό επίπεδο και τα, οι πόροι για την Ήπεθρο θα πρέπει να υπόψη, να συντονίζονται με τα διάφορα εδαφικά μέσα της συνοχής. Το ΑΕΠ Άκουσα αυτά που είπε και ο Σπίπερ προσεκτικά για τα μέτρα μετά το ΑΕΠ όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις ή την εθνική ευμάρεια. Το ΑΕΠ θα πρέπει να είναι βασικό στοιχείο αναφοράς. Βασικό κριτήριο για την επιλεξιμότητα. Και μπορούμε εύκολα να αξιολογήσουμε τι θα ακολουθήσει το 2013 και να βρούμε τα κατάλληλα μέσα. Συνεργαζόμαστε πολύ καλά με τον Ιωάννη Χάν. Να κινηθούμε σε ευρύ ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο σε εκείνους που δικαιούνται βοήθεια από το στόχο 1 ή στόχο 2 της πολιτικής συνοχής. Θέλουμε απλούστευση. Η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού ήδη είναι στα χέρια της Ίγκε Γκρέσλερ. Δύσκολο αυτό για μένα. Ήδη ηγείται όμως εκείνη στον τομέα με ανεκτό επίπεδο ποσοστό κινδύνου. Έχουμε αυτό τον όρο, αυτή την έννοια στο δημοσιονομικό κανονισμό. Και έχουμε καλά νέα όσον αφορά το πραγματικό επίπεδο σφάλματος στην πολιτική συνοχής. Θέλουμε να δούμε τι δυνατότητε έχει ο ευρωπαϊκό προπολογισμό και να στηρίξουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό μέσω καινοτόμων μέσων, προγραμμάτων ε, επιμερισμού του κινδύνου συνεργασία ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο δημοσιονομικό κανονισμό και στη θετική αναθεώρηση. Και τέλο, κάτι εξίσου σημαντικό, να απαντήσουμε στο εξή ερώτημα. Πέρα από τι μεγάλε αστικέ περιοχέ που σωρεύουν προβλήματα, πώς να συμπεριλάβουμε τις μακροπεριφέρειες, αυτή την έννοια. Βαλτική, Μεσόγειος, Εύξηνος Πόντος στο μελλοντικό όραμα για την περιφερειακή πολιτική. Αυτό που προσοσήτηση. Ο Ιωάννης Χάν δεν είναι θερμός υποστηρικτής αυτού ξεχωριστών δομών για μάκρο περιοχές. Θέλει ολοκληρωμένη περιφερειακή πολιτική με κάποιες περιφερειακά μακρό μορφώματα. Αυτές είναι κάποιες υποθέσεις για το μέλλον. Αυτό που έχει σημασία είναι η συνοχή να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο των συζητήσεων για το μέλλον των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Υπάρχει κλίμα απογοήτευσης, κλίμα λιτότητας, προγράμματα λιτότητας. Επηρεάζουν αρνητικά την κατάσταση. Πώς το χρέος επηρεάζει τη συγχρηματοδότηση, τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης των Ομοσπόνδων Κρατηδίων της Γερμανίας, πραγματοσχάρη. χάρη. Όλα αυτά πρέπει να εξεταστούν, να εξολογηθούν. για να καθορίσουμε στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο την πολιτική της συνοχής. Αυτά εν γέννη και θέλω να ακούσω τις απόψεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μεγάλο κατάλογο αγορητών. Μετά από τρεις αγορητές θα δίνουμε το λόγο στον Επίτροπο. Ο κύριος Βόντ είναι ο πρώτος. I don't, I, I have Mr. Uh, on the list. Yeah. I think that's me. Oh. Uh, Νομίζω ότι εννοείται εμένα. Θα είχα πολλά να πω για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε εδώ και για την ε, πολιτική συνοχή και για τα εθνικά ταμεία. Αλλά τώρα θα ήθελα να επικεντρωθώ στο σημερινό ζήτημα. Και καταλαβαίνω γιατί τα κράτη-μέλη επιφυλάσσονται αυτή τη στιγμή στις περικοπές που γίνονται όπως θεωρούν κατά των ίδιων των χωρών τους ή δεν θέλουν να αυξήσουν τις συνεισφορές τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η συνθήκη της Λισαβόνας, οι νέε ευθύνε, η ίδρυση μιας υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, οι πρωτοβουλίες για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Νομίζω ως πρώην μέλος της Επιτροπής Προπολογισμού καταλαβαίνετε τώρα τι νέες μεγάλες πιέσεις ασκούνται στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό ακριβώς εξαιτία αυτών των νέων ευθυνών. Τα πράγματα λοιπόν ε, γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Και νομίζω ότι θα ήταν σφάλμα η, τα κονδύλια στο 1α και 1β να περιοριστούν. Εδώ θα πληγούν οι, οι επενδύσεις. Και οι επενδύσεις μακροπρόθεσμα και για σκοπούς ανάκαμψης πρέπει να είναι ελεύθερες και για τον 2011 ε, θα υπάρχει η προοπτική περικοπή στο 1α 46 εκατομμύρια και 891 εκατομμύρια στις πληρωμές. Θα πρέπει όμως να μην ξεχάσουμε ότι το 1α προσφέρει σημαντική χρηματοδότηση για όλες τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κόστο λοιπόν θα πρέπει να το καλύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε πώ θα μεταφερθεί το κόστο και πώ θα συνδυαστεί με το 1β. Θα πρέπει τα ερχόμενα χρόνια να δούμε πώς μπορούν να, να αντισταθμιστούν αυτά τα δύο. Νομίζω εδώ ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάποιε τεχνικέ διευθετήσεις στο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο αντί να βρούμε πραγματικέ λύσει. Εσεί Είστε πρόθυμος να εξέβρετε τέτοιες πραγματικές λύσεις και να δείτε τι θα γίνει με τις κατηγορίες 1α και 1β, ώστε μακροπρόθεσμα να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη ανάκαμψη οικονομική στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Σωστά αναφερθήκατε στην ένταση που υπάρχει μεταξύ διαφορετικών πολιτικών ε, κατευθύνσεων και των ε, χρηματοδοτήσεων τους επίσης. Δηλαδή πολλά κράτη-μέλη θέλουν να εξασφαλίσουν μια παγιοποίηση του προϋπολογισμού τους, μια εξυγίανση του προϋπολογισμού τους που θα έχει και κάποια συνέπεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα είναι πώς θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι τέτοιο. Το δεύτερο ερώτημα συνάπτεται με τη ζώνη του ευρώ. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολύ λίγα εργαλεία τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στη μακροοικονομική σταθεροποίηση και από την πλευρά της Κομισιόν δεν έχω ακούσει πολλά για το αν σκέφτονται στο μέλλον να ενισχύσουν το, την μακροοικονομική σταθεροποίηση στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας και το Ταμείο Συνοχής. Εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω ή να επικρίνω τον Επίτροπο τον κύριο Ρέεν, αλλά θα ήταν πραγματικά αντιπαραγωγικό να αποκοπούν τα Ταμεία Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία για χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα, ενώ πράγματι θα πρέπει στις χώρες αυτές να λάβει η χώρα μια μακροοικονομική σταθεροποίηση. Και πολλές φορές για τις χώρες αυτές είναι χώρες, πρόκειται για χώρες που έχουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας και τα ταμεία συνοχή και τα διορθωτικά ταμεία έχουν σημαντικό ρόλο για να μπορέσουν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των χωρών αυτών. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η άποψή σα για το θέμα αυτό. Τέλο, μια πάρα πολύ σύντομη ερώτηση. Πώ γίνεται ο πρόεδρο Μπαρόσο να βρει ξαφνικά, να έχει βρει ξαφνικά ένα δισεκατομμύρια ευρώ που υποσχέθηκε στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για στόχους ανάπτυξης Μήπως πρόκειται για χρήματα τα οποία δεν θα εκταμιευθούν από την πολιτική συνοχής, εν μέρη τουλάχιστον. Thank ε, Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την εξαιρετική του εισήγηση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει στενή σχέση συνεργασία μεταξύ Επιτροπή και προπολογισμού για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Όπω είπατε, ο προπολογισμό θα είναι πολύ σκητό για το επόμενο πολιτέ πλαίσιο. Και η όλη συζήτηση για του ιδίου πόρου θα επηρεάσει ιδιαίτερω την εξέλιξή του. Νομίζω λοιπόν είναι σημαντικό να εξετάσουμε ποιε είναι οι προοπτικές για τι διάφορε συναλλαγέ και αλλαγέ που πρέπει να επιφερθούν στη φορολογική πολιτική λόγου χάρη. Εγώ είμαι κάπω επιφυλακτική όταν μιλάμε για πέντε προοπτικέ σε βάση πενταετία. Λόγω χάρη για τα διευθυντικά ταμεία, πώ θα τι ε, προσαρμόσουμε στο επίπεδο τη πενταετία. Και αυτό που λιγάκι με εκνευρίζει και με ενοχλεί είναι ότι αφότου έχω συμμετάσχει στη συζήτηση περί προπολογισμού και έχει ακουστεί και το θέμα του πόσο άκαμπτος έχει γίνει πλέον ο προπολογισμό και πώ θα πρέπει να προσαρμοστούν οι παραδοσιακέ πολιτικές και να συνδυαστούν με τις νέε, η δική μου απορία είναι εξή. Ποια θα είναι η σχέση με τις νέε αυτέ πολιτικές. Φαίνεται να μην υπάρχει, γιατί συνήθω μιλάμε διαρκώς για αλληλεγγύη, για βοήθεια και υποστήριξη, αλλά δεν μπορούμε να διαδούμε ποιε είναι οι δυνατότητε που ανοίγονται μπροστά μα και όσο σε ό,τι αφορά τη στρατηγική τη Ευρώπη του 2020, εδώ πρέπει να αναζητήσουμε την προστεθέμενη αξία και για την πολιτική τη συνοχή. Θα πρέπει εμεί να προσφέρουμε τη στήριξή μα για του διάφορου στόχου μα, όπω τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, τι πράσινε πολιτικέ. Οι πόροι και οι δυνατότητε που προσφέρουν για συγκεκριμένε περιφέρειες και περιοχέ είναι πολύ σημαντικοί. Έχουμε παραμελήσει λοιπόν την συζήτηση αυτή και τη διασύνδεση των παραδοσιακών πολιτικών με τις νέες. Θα πρέπει λοιπόν νομίζω να έχουμε μια θεώρηση πιο ευρεία του όλου θέματος. Επίση, θα πρέπει να ενισχύσουμε την πολιτική συνοχή και να αναζητήσουμε νέες προτεραιότητες λόγω χάρη στην έρευνα, να μια από τι πρώτε προτεραιότητε που θα έπρεπε να θέσουμε. Ελπίζω ότι όλα αυτά θα τα λάβετε υπόψη στι μελλοντικέ σα συζητήσει Και σε ό,τι αφορά τα κριτήρια, να πω πολύ σύντομα ότι συμφωνώ απόλύτω μαζί σα, ότι το ΕΠ θα πρέπει να είναι ένα από τα πρωταρχικά κριτήρια, αλλά θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και με τι μελλοντικέ προκλήσει. Η γύραση του πληθυσμού, λόγω χάρη. Πώ θα μπορέσει η πολιτική συνοχή να ανταποκριθεί σε αυτέ τι νέε προκλήσει. Και έπειτα θα ήθελα, ολοκληρώνοντα, να ζητήσω και τη γνώμη σα για την πολιτική των μεταφορών. Έχουν γίνει συζητήσει σχετικά και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Κάλλας, ε, ανέφερε ήδη κάποιες ιδέες όπως λόγου χάρη να δημιουργηθεί ένα ίδιο ταμείο για ε, το θέμα της, ε, των μεταφορών. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Thank you. This the Σας ευχαριστώ. Πήρα μια γεύση των μελλοντικών συζητήσεων. Δεν είναι τόσο εύκολε οι ερωτήσει από την αρχή. Για τον κύριο Βον, δεν ξέρω αν προφέρω σωστά το όνομα σα. Α, κοντά, ε. Εντάξει, ευχαριστώ για την ανοχή σα. Ξέρω ήδη ότι με τη λογική μας της αναθεώρησης είμαστε υπολοιπόμεθα των προσδοκιών του Κοινοβουλίου. Θέλαμε να ευθυγραμμιστούμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας χωρίς να τροποποιήσουμε περισσότερο τα πράγματα από όσο απαιτεί η νέα συνθήκη. Το Κοινοβούλιο, και αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση του συναδέλφου Ράιμερ Μπέγκε, είναι να γίνει πιο πολιτική προσέγγιση στο θέμα, όχι ευθυγράμμιση απλώς στην συνθήκη της Λισαβόνας. Ποιο είναι το πρόβλημα. Κάτι που θα ξεκαθαριστεί αύριο, στην Κομπού που ψηφίζει τροπολογία στην έκθεσή του. Εκεί θα δούμε τι συγκεκριμένο θα γίνει. Μη ευθυγράμμιση τη Λισαβόνα, αλλά πλέον πολιτική συζήτηση αναθεώρηση. Χωρί νομική βάση δεν μπορούμε να αποσωτικοποιήσουμε τι νέε ευθύνε απορρέουν από τη Λισαβόνα. Υπάρχουν νέε ευθύνε σε πολλού τομεί, αλλά χρειάζεται νομική βάση για να μπορέσουμε να αποσωτικοποιήσουμε τι ευθύνε αυτέ. Είμαστε με την ευθυγράμμιση εμεί και υπολοιπόμεθα των προσδοκιών του Κοινοβουλίου. Αυτό που είναι σίγουρα ορατό στις τροπολογίες του προπολογισμού του 2010 είναι η υπηρεσία εξωτερική δράσης. Με το διορθωτικό προπολογισμό μέχρι 9,5 εκατομμύρια ευρώ και νέες γραμμές και νέες θέσει. αυτό δεν είναι κάτι δημοφιλέ προ του Ευρωπαίους, η αύξηση των διοικητικών δαπανών. Αλλά αυτή είναι θέμα τη ορατότητα τη Λισαβόνα, εξωτερική δράση. Κάτι που θα αναπτυχθεί και θα ληφθεί υπόψη και στο μέλλον. Όσον αφορά αθλητισμό και πολιτισμικά, είναι η στρατηγική του Κοινοβουλίου για τι διαπραγματεύσει του 2011 και θεωρώ ότι είναι εφικτή η προσπάθεια για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Θα φαίνεται και στον προβλησμό του 2011. Βλέπω σχετικές Συγκεκριμένε τροπολογίε του εισηγητού για τον προπολογισμό. Προσελκύσατε την προσοχή μα στι περικοπέ. που είναι πολύ μεγάλε στο κεφάλαιο 1, κατηγορία 1, στην 1α και στην 1β. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο μεταξύ λόγων και πράξεων. Όλοι λένε ότι η Ευρώπη πρέπει να δαπανά περισσότερη ανταγωνιστικότητα για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της αλλά όπως είδαμε και σε 2005 2005-2006, εδώ έγιναν οι μεγαλύτερες περικοπές. Οι πολιτικοί υπερασπίστηκαν λιγότερο αυτό το κομμάτι του προϋπολογισμού και έγιναν οι περικοπές παρά τις δηλώσεις περί ανάγκης επενδύσεων στην ανταγωνιστική Ευρώπη και την έρευνα. Το ίδιο ισχύει τώρα και με τις περικοπές που θέσπισε το Συμβούλιο. Επικεντρωθήκαμε κατά 96% των αυξήσεων 2011, εν συγκρίση το 2010, στο 1α και 1β. Αυτό που θα έπρεπε κανονικά ένα καλό μήνυμα ποιο είναι η πρόθεση της συνοχής. Το 2010 ένα δις παραπάνω έπρεπε να ξοδευτούν από αυτά που είχαν προγραμματιστεί στον προϋπολογισμό για το 2011, δις παραπάνω. Διότι όλοι τώρα προχωράνε για να καλύψουν καθυστερήσει. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και το 2011, 2012, 2013. Αυτού του είδου τις δαπάνε εγώ τις υποστηρίζω, διότι είναι στα πλαίσια των επενδύσεων. Και είναι μικρά προγράμματα καταπολέμησης τη κρίσεω που επηρεάζουν και τις θέσει εργασία και τη συνεργασία θετικά. Είναι κάτι καλό. κάνουμε τη σύγκριση. Ε, ανάκαμψη, λιτότητα, τι θα ακολουθήσουμε. Ακολουθούν διαφορετικές προσοχές στα κάτι μέλη. Τα, το θέμα των επενδύσεων πρέπει να συζητηθεί. Και σε περίοδο λιτότητας. τι γίνεται. Έχουν γίνει σοβαρές περικοπές σε επενδύσει στην Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία και σε άλλε χώρε. Θα μπορούσαμε να καλύψουμε το κενό μέσω διεθντικών ταμείων που κανονικά αφορούν επενδυτικούς πόρους με πολλαπλασιατικό αποτέλεσμα. Αυτά λέω είναι ήδη απαντήσω στον κύριο Τόρερ. Στο ερώτημα δηλώ, ε, λιτότητα έναντι ανάκαμψης. Μπορούμε με τα μέτρια μας αυτά μέσα να συμβάλλουμε στη σωστή λύση. Δεν ξέρω πού μπορούν να βρεθούν τα ένα δις για την ανάπτυξη. Αλλά είμαστε τόσο δημιουργικοί στη συνδιαλλαγή και ίσως μπορέσουμε να βρούμε χρήματα για επισητιστική βοήθεια, για το Γαλιλαίος, για προγράμματα ανάκαμψης. Χρειαζόμαστε ευελιξία, βλέπετε, και πρέπει να την υπερασπιστούμε την ευελιξία. Ευελιξία στα πολιτή προγράμματα. Κυρία Μάνερ, δεν θέλω να αναφερθώ στη φορολόγηση πολύ. Θα προστιμούσα να αναφερθώ στους ιδίους πόρους, σύμφωνα με τη συνθήκη, και όχι η φορολόγηση. Η φορολόγηση δημιουργεί τρόμο. Θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια να μειώσουμε την εθνική συνεισφορά για να βοηθήσουμε τους υπουργού Οικονομικών. Στη διαδικασία αυτή, στήριξη των οικονομικών. Ε, επίσημα κατακρίνουν, ανεπίσημα υποστηρίζουν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ψάχνουν να βρουν τις δυνατότητες να μειώσουν την εθνική συνεισφορά, ούτω ώστε να διευκολύνουν τη ζωή τους όσον αφορά την στήριξη των δημοσιονομικών. Ό,τι προτείνεται, είτε, ε, είτε φορολόγηση χρηματοστικών συναλλαγών είτε οτιδήποτε άλλο, το βλέπουν σαν εθνικό εισόδημα να μην το μοιραστούν με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Προσπαθούν απελπισμένα να βρουν και άλλε πηγέ εσόδων σε εθνικό επίπεδο, όχι ευρωπαϊκό. Άρα είμαι αρκετά διστακτικό, αλλά είμαι υποχρεωμένο να παρουσιάσω τι επιλογέ με τον, περισσότερο, με τον πιο ουδέτερο τρόπο. Συμφωνώ μαζί σας κυρία Μάνερ ότι πέντε χρόνια θα δημιουργήσουν ξανά νέα διαμάχη για νέους πόρους. Θα δούμε τι θα γίνει τον επόμενο χρόνο. Δεν θέλουμε διαμάχες γιατί αυτές χωρίζουν την Ευρώπη, δεν ενώνουν την Ευρώπη. Όταν δημιουργούνται επίμαχα θέματα, σε πέντε χρόνια θα μπούμε σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων. Μετά από δύο χρόνια, για την νέα πενταετία, επί της βάσεως των αρχικών δημοσιονομικών προοπτικών, Τα πρώτα δύο χρόνια δεν δείχνουν δώσει αποτελέσματα. Τον τρίτο χρόνο, τον τέταρτο χρόνο φαίνονται τα αποτελέσματα του προγραμματισμού περισσότερο. Εγώ δεν είμαι πρόμα, ε, υπέρμαχος της πενταετίας. Μετά από μία δοκιμή στις πρώτες δημοσιονομικές προοπτικές επέλεξα αυτή τη θέση. Ο Ράιμον Μπέγκε έλεγε ότι θα έπρεπε να προσαρμόσουμε την εντολή που δίνεται στο Κοινοβούλιο. Εγώ προτείνω να επεκταθεί η θητεία του Κοινοβουλίου μάλλον σε, πέντε χρο... σε 7 χρόνια. Δεν ελήφθη υπόψη αυτή η πρόταση, δεν έγινε αυτή η προσαρμογή για κάποιους λόγους. 2012-2020. Η προσαρμογή είναι κάπως τεχνητή σε αυτή τη δομή. Εντοπίζουμε απλώς τις δαπάνες που οδηγούν σε πράσινη ευφυή ανάπτυξη. Αντί να αναπτύσσουμε διάφορες κατηγορίες δαπανών. Στο μέλλον, ευθυγραμμίσει με τη φιλοσοφία του 2020 θα πρέπει να είναι κάτι που λαμβάνεται υπόψη στον προσανατολισμό του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Είπε σαφώ ότι είμαι υπέρ ολοκληρωμένη ε, πολιτική συνοχή. Υπάρχουν τρει τομεί όπου γίνεται προσπάθεια για ανεξαρτησία πέρα από το κοινωνικό ταμείο. Καταρχήν έχουμε τις μεταφορές για τα ευρωπαϊκά δίκτυα, δεύτερον έχουμε τον τομέα της ενέργειας και τρίτον του κλίματος. Εγώ θέλω να υπερασπιστώ μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να βρούμε χρήματα τα οποία θα υποστηρίξουν την εδαφική συνοχή και δεν θα οδηγήσουν σε κατακαιρματισμό σε πάρα πολλά ταμεία. Γιατί αυτό σημαίνει και αύξηση του διοικητικού άχθους και του διοικητικού κόστους αν έχουμε ανεξάρτητους φορείς, όλοι αυτοί οι αυτόνομοι ανεξάρτητοι φορείς χρειάζονται <clears throat> ανεξάρτητα, ανεξάρτητες διοικήσεις και το ε, συμπαρομαρτούν διοικητικό κόστος. Αλλά δεν είναι εύκολο να το αποφύγουμε πάντα. Ο πιο εύκολος τρόπος να υποσκάψουμε όχι τον προϋπολογισμό, μονάχα αλλά και την ε, αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διονγκώνοντας τον ε, διοικητικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι αυτό κοιτάνε στην Ευρώπη. Ε, δεν είναι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού, αλλά αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να υποσκάψει την αξιοπιστία της Ευρώπης, το να έχουμε μεγάλο διοικητικό προϋπολογισμό. Ο Τζον Μπάρτον έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γεια σας κύριε Επίτροπε την προηγούμενη εβδομάδα 7 δημοτικά συμβούλια στην Ανατολική Ουαλία συζήτησαν για την Ευρώπη του 2013 και επέκεινα και κατέληξαν σε μία δήλωση. Έχουν κανονικά ε, διεκδίκηση 110.000 ε, από διάφορα προγράμματα περιφερειακά και επίσης και άλλες ε, Δυνατότητε χρηματοδότησης. Με την αλλαγή των δημοσιονομικών προοπτικών θα υπάρξει επίπτωση σε πολλά ε, σχέδια με μεγάλη επίπτωση και στην απασχόληση. 15 που είναι περιφερειακού χαρακτήρα, 8 τα οποία είναι ε, απασχόλησης και 16 για στρατηγικού στόχου. Όλα αυτά λοιπόν εξαρτώνται από τη συνέχιση της χρηματοδότησης για τα θέματα αυτά. 6% μονάχα είναι τα χρήματα που δίνονται για, του προπολογισμού μόνο για απασχόληση. Και αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει να το συγκρίνουμε με το 1 δισεκατομμύριο που έχουμε υποσχεθεί στην Ελλάδα και άλλες χώρες για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του προπολογισμού τους. Οι αλλαγέ στον προπολογισμό θα οδηγήσουν σε μεγάλα προβλήματα στην Ουαλία, όπου η απώλεια τη μεταπηδική βιομηχανία έχει οδηγήσει σε μαύρη τρύπα απασχόληση. Αυτέ οι θέσει απασχόληση βρίσκονται στο στόχαστρο η μείωση της χρηματοδότησης θα οδηγήσει ακόμα μεγαλύτερη αθλειότητα στην Ουαλία που έχει το υψηλότερο επίπεδο ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό σημαίνει όλο και αυξανόμενο κόστος του να ανήκει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν τα χρήματα αυτά χρειάζονται για τις περιοχές μας. Δεν είμαι έτοιμος να αποδεχτώ μια ελαφρά την καρδία κατάργηση κονδυλίων τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωση της Ουαλίας. Δεν καταλαβαίνω γιατί στέλνουμε, δίνουμε λεφτά σε μια χώρα η οποία έχει ήδη οικονομικά προβλήματα και υψηλή ανεργία. Αν αυτό τώρα ευθυγραμμίζεται με το στόχο της Ευρώπης του 2020, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Θα πρέπει να υπάρξει μια αξιολόγηση από την Κομισιόν για να καταγραφούν οι αρνητικές συνέπειες της απόσυρσης της υποστήριξης προς περιοχές όπως η Ουαλία που κινδυνεύουν να πέσουν σε βαθιά ύφεση. Μπορείτε να εξετάσετε λοιπόν την αίτησή μου. Η κυρία Μανέσκου. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε για την ε, παρουσίασή σας. Θα ήθελα να σας πω ότι με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω ότι συμμερίζεστε κατά τη δική μου την άποψη θα στηρίξετε τι αρχέ τοπική αυτοδιοίκηση και περιφερειακή αυτοδιοίκηση μέσω τη πολιτική συνοχή, λέτε. Αυτό λοιπόν με ικανοποιεί ιδιαίτερα. Ελπίζω ότι θα υποφεληθούμε τη στήριξή σα. Και εφόσον εκφράσατε αυτήν σας την προοπτική στήριξη των ε, περιφερειών και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, να σας πω ότι θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην ε, κατάρτιση και την εκπαίδευση των ε, λειτουργών και υπαλλήλων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Διότι εκείνοι άμεσα εμπλέκονται στην ε, υλοποίηση των προγραμμάτων των διευθυντικών ταμείων και της πολιτικής συνοχής. Πιστεύετε λοιπόν ότι μέσω της Επιτροπής της ίδιας μπορεί να υποστηριχθεί ένα πρόγραμμα ή να προταθεί ε, ένα πρόγραμμα που να διευκολύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών ε, μεταξύ των ε, εργαζομένων στις διάφορες τοπικές ε, περιφερειακές αρχές. Ένα πρόγραμμα για τη μόρφωσή τους δηλαδή και για να βελτιώσουμε την διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Να έχουμε μια αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτών των ταμείων. Ένα άλλο τώρα ερώτημα σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής, εφόσον είναι ένας παράγων ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να συμβαδίζει άλλωστε και με την στρατηγική του 2020. Η πολιτική συνοχής δεν είναι πολιτική φιλανθρωπίας. Δεν έγκυται απλά στην αλληλεγγύη, αλλά και στην ανάπτυξη, την ε, συνεκτική και αποτελεσματική ανάπτυξη των διαφορών περιφερειών, ώστε να απαλληθούν μεταξύ τους ανισότητες. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποια είναι η δική σας η άποψη σε σχέση με το μέλλον της πολιτικής συνοχής από την προοπτική του προπολογισμού. Θα πρέπει να διατηρήσουμε το ίδιο δημοσιονομικό πλαίσιο Θα πρέπει να, δια, να διατηρήσουμε ανέπαφε στις αρχές και τα ποσά που αποδίδονται στην πολιτική συνοχή ή εσείς έχετε μια διαφορετική θεώρηση και αν ναι, είναι αυτή. Ευχαριστούμε. Ο, η κυρία Μανέσκου είναι συντονίστρια για την ομάδα Άλντε και τώρα συντονίστρια των Χριστών Δημοκρατών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι εξαιρετικό το ότι μπορώ να σας υποδεχθώ στην Επιτροπή μας θυμάμαι την ε, συνεργασία που είχαμε και στο παρελθόν και είναι σημαντικό το θέμα αυτό για την προετοιμασία της πολιτικής συνοχής στο μέλλον. Εγώ έχω ορισμένα ερωτήματα να σας θέσω. Εγώ δεν θεωρώ ότι οι κυρώσεις θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν από την τωρινή του οικονομική πολιτική σε μια πολιτική που ευνοεί τη συνοχή. Νομίζω ότι είναι λανθασμένη μια τέτοια προσήγηση, αλλά το ερώτημα είναι εσείς σκέφτεστε και άλλα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Γιατί η πολιτική συνοχής είναι ένα σημαντικό στοιχείο μέσα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. που υπάρχουν λοιπόν άλλα μέτρα τα οποία μπορεί να επιβάλλει κανείς και όχι να αποκόψει τα ποσά του Ταμείου Συνοχής. Αναφερθήκατε δεύτερον στο, στα ταμεία για τις μεταφορές φοβάμαι ότι υπάρχει μια όλο και μεγαλύτερη αντιμετώπιση κατατομής της πολιτικής μεταφορών και επομένως και αυτό γίνεται ε, αιτία να υπάρξουν ανταγωνισμοί μεταξύ των διαφόρων τομέων. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά, το Ταμείο για τα, η πολιτική για το, τις μεταφορές, για την ενέργεια, για την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά πρέπει να βρουν κάπου πόρους και κατατρώγουν πόρους της πολιτικής ε, συνοχής. Εσείς πιστεύετε ότι είναι σωστή αυτή η αντιμετώπιση κατά το ή μήπως η Κομισιόν σαν συλλογικό σώμα θα πρέπει κάποτε να μπορεί να λέει και όχι σε τέτοια κατάτμιση των πολιτικών και των ε, κονδυλίων. Τρίτον, νομίζω ότι μέσα στην Επιτροπή μας έχουμε μία γενική συνένεση ότι ο χρόνος διάρκειας των προοπτικών αυτών θα πρέπει να είναι πράγματι 7 χρόνια. Ο πρώτος Μπαρόσο είχε θέσει τη δυνατότητα να είναι και μικρότερη η, η διάρκεια αυτών των προοπτικών. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ένα χρονικό διάστημα το οποίο θα είναι επαρκές για να μπορούμε να προγραμματίσουμε σε σωστό επίπεδο, αλλά αρκετά σύντομο συγχρόνο χρόνο για να μπορούμε να αντιδρούμε ταχαίω όταν χρειάζονται αλλαγέ. Ποια είναι η άποψή σε σχέση με τι χρονικέ διάρκειε των προγραμμάτων από την Κομισιόν. Ο κύριο Επίτροπο έχει το λόγο. Κύριε Μπάρτον, είναι πολύ σκληρό το επιχείρημα σα υπέρ τη πολιτική συνοχή και τη περιφερειακή πολιτική και μάλιστα με βάση τι εμπειρίε τη Ουαλία. Βεβαίω, τη γενικότερη εικόνα του μέλλοντο των περιφερειών τη Μεγάλη Βρετανία πρέπει όλα αυτά να λαμβάνονται υπόψη. Τώρα για την επιλεξιμότητα των ε, συγκεκριμένων ε, επαρχιών μεταξύ των 271 ε, που υπάρχουν στην Ευρώπη. Θα ακολουθήσουμε μια σαφή μεθοδολογία. Και όπως είπε και η κυρία Μανέσκου, δεν αρκεί για το μέλλον να έχουμε πλήρη στήριξη υπέρ της συνοχής μόνον, αλλά θα πρέπει να παραμείνουμε ακριβώς πιστοί σε αυτή τη μεθοδολογία, τη μεθοδολογία του Βερολίνου. Δηλαδή, εκτός από τους ε, στόχους υπαριθμών 1 της πολιτικής συνοχής και τους υπαριθμών 2 και τις ε, πολιτικές που εφαρμόζονται σταδιακά στις διάφορες περιοχές κατά ε, ανωδικά ή μειωτικά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ποσοστό και τα αστικά κέντρα. Και να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες της κάθε περιφέρειας, όπως στην περίπτωση της Ουαλίας. Και το θέμα είναι πώς θα κερδίσουμε ευρωπαϊκή στήριξη για την πολιτική συνοχή. Υπάρχει λοιπόν η μεθοδολογία του Βερολίνου, αλλά υπάρχουν και δύο προσαρμογές. Προκειμένου να μην χάσουμε τη στήριξη της Ισπανίας, και της, τη συμφωνία της ε, Γερμανίας. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το μέρος, το θέμα της Ανατολικής Γερμανίας, της Προανατολικής Γερμανίας, της Έστιλαντ. Παντώ σίγουρα θέλουμε να φέρουμε του ανθρώπου με το μέρο τη πολιτική συνοχή και τη περιφερειακή πολιτική. Για να πετύχουμε συμφωνία το 2012, πρέπει να σκεφτούμε ότι κανεί δεν θέλουμε να βγαίνει χαμένο από την εικόνα που θα διαμορφωθεί στο μέλλον. Για να υπάρξει συμφωνία μεταξύ 27 κρατών, δεν μπορούμε, κανείς να, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κανεί να χάσει μεγάλα πλεονεκτήματα. Θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε μια προσφορά ενδιαφέρουσα και δελεαστική για όλους. Η βασική λοιπόν συνέπεια της αρχικής μας φιλοσοφίας είναι ότι δεν θέλουμε να έχουμε μεγάλους χαμένους σε όλες αυτές τις διαρροματεύσει. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε κάτι λοιπόν και για την περιοχή που σας είναι τόσο προσφυλής. Αλλά για να απαντήσω τώρα και στην κυρία Μανέσκου, δεν αρκεί η μεθοδολογία του, του Βερολίνου, όσο και αν είναι θεμελιώδης αρχή μας. Θα πρέπει Σίγουρα σε αυτή να βασιστούμε, αλλά θα χρειαστούν και προσαρμογές για τα αστικά κέντρα, λόγου χάρη, την συσσόρευση μεγάλων προβλημάτων εκεί. Θα πρέπει εκεί να αναζητήσουμε συγκεκριμένες λύσεις για τα μεγάλα αστικά κέντρα, για να τις φέρουμε και αυτές με τη δική μας την πλευρά την πλευρά υποστήριξη τη περιφερειακή πολιτική δηλαδή. Και αυτό είναι και ένα γεγονό αναντήρητο τη καθημερινότητα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα θα υπάρχει σώρευση πραγματικών προβλημάτων που θα πρέπει να λυθούν και με την μετριασμένη αυτή συμβολή του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Σίγουρα υπάρχουν ήδη προβλεπόμενες δυσκολίες με τις μελλοντικέ μας προτάσεις, όμως υπάρχουν και εξελίξεις θετικές. Ε, Ω τώρα στι προηγούμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ είχαμε 16-17% ένα μερίδιο για την ε, πολιτική συνοχή, τώρα φτάνουμε το 36%. Ε, μπορούμε να φτάσουμε στα επίπεδα της γεωργίας. όχι. Δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια επαναστατική προσέγγιση και εκεί στα αγροτικά. Θα πρέπει κάθε χώρα να στηρίξει με δικά της κονδύλια τις φιλοδοξίες έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν θέλω τώρα να προδικάσω αυτή τη συζήτηση. Έχω δεχτεί ειδική πρόσκληση και από την Επιτροπή Γεωργίας και θα φροντίσω εκεί να τα σχολιάσω αυτά. Πάντως, για να αποσαφενιστεί ο ευρωπαϊκός Προπολογισμό, πρέπει να βρούμε λογικές προτάσεις. Προτάσεις ε, ορθές λογικές για να υπάρξει χρηστή χρήση του προπολογισμού. Και βεβαίως να είναι και θεμητοί οι στόχοι που θέτουμε, κάτι που είναι σημαντικό για το πώς δαπανώνται τα κονδύλια ε, στον 21ο αιώνα πια. Κυρία Κρέλ, για τις κυρώσεις δεν είναι ακόμη τόσο σαφές ποια διευθυντικά μέτρα πρέπει να προληφθούν. Για το άρθρο 136 της συνθήκης της Λισαβόνας νομίζω είναι λιγότερο επίμαχο ε, από ότι γενικότερα εκτός Ευρωζώνης. Ισχύει λοιπόν πιο πολύ για την Ευρωζώνη, αλλά εδώ μας ενδιαφέρουν οι 27 χώρες, όχι μόνο αυτές της Ευρωζώνης. Και πρέπει να ανατρέξουμε και στον προπολογισμό, αλλά με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα. Γιατί εάν υπάρχουν συνθήκες ύφεση και στερούμε από τα μη πειθαρχημένα προ... κράτη-μέλη με προβλήματα λιτότητας, σφιχτών δημοσιονομικών. Τα στερούμε λοιπόν από δυνατότητες για το μέλλον. Αυτό δεν μπορεί να επιτραπεί. Και δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι αμέσως. Δεν μπορούμε να, να στείλουμε τις δεσμεύσεις μας για δύο χρόνια, να περιοριστούν οι πληρωμές, να υπάρξουν περικοπές στις πληρωμές και για την πολιτική συνοχή. Αυτό μπορεί να γίνει αλλά μετά από μία περίοδο μεταβατική. Πρέπει να υπάρξει μια ευελιξία. Οι ενδεχόμενες κυρώσεις πρέπει να τεθούν και να προβλεφθούν με τρόπο ε, ήπιο, ώστε να μην υποβαθμιστεί η, περαιτέρω η οικονομία μιας συγκεκριμένης χώρας. Νομίζω αυτό το απήντησα και στην προηγούμενη ομάδα ερωτήσεων. Πάντως, θα πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από την όλη κρίση. Χρειάζονται κάποια εργαλεία και προληπτικά και διορθωτικά και σίγουρα πρέπει να, τα, να σκεφτούμε πώς θα τα σχεδιάσουμε αυτά. Νομίζω βέβαια υπάρχουν και άλλες τάσεις, γερμανικές ίσως να πάμε ακόμη πιο μακριά, αλλά το θέμα είναι να δούμε πώς θα επιβάλλουμε καιρό σε μια συγκεκριμένη περιοχή, που να είναι και ορατές, αλλά να μην πλήξουμε περαιτέρω αυτή την περιοχή. Και έχω πει επανειλημμένω στην Επιτροπή ότι είμαι ενάντια στην αποσταθεροποίηση και την τομεακή, αυστηρά τομεακή προσέγγιση στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αυτό και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι στην πολιτική του 2020, αλλά χρειάζονται και κάποια εχέγγυα για το ταμείο αυτό, προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Στην πολιτική μεταφορών πάντως μπορούμε να βρούμε κάποιες λύσεις ε, και με την πολιτική συνοχή. Για την επταετία τώρα, αυτή είναι η δική μου η προτίμηση. Μετά την πενταετία θα πρέπει να υπάρξει μια πραγματική αναθεώρηση. Θα μπορούσα να συμφωνήσω με το 5 συν 5, αρκεί να υπήρχε αναθεώρηση στο μέσον, αλλά αναθεώρηση σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και κάποιο ε, δυναμικό, για το, κάποιο ενεργητικό για το μέλλον διότι αναθεώρηση σημαίνει ακριβώς αυτό, αποθεματικό. Μια θεωρητική αναθεώρηση που δεν μπορεί να οδηγήσει και σε επανεξέταση δεν έχει νόημα. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να δούμε τις δημοσιονομικές προοπτικές ε, και το κλίμα αυτό που υπάρχει για το ευρώ, αλλά όχι μόνο στην απεσιόδοξη πλευρά του, θα παγώσουν τα πράγματα για μια δεκαετία. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τώρα καθορίζουμε το κλίμα για το μέλλον. Δεν πρέπει να είμαστε μόνο απεσιόδοξοι. Θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και σίγουρα η δική μου προτίμηση είναι το 5 συν 5. Ε, Συνάδελφοι, έχουμε 7 που θέλουν να μιλήσουν σε ένα 20 λεπτό. Παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι και ο Επίτροπος το ίδιο. Για Κυρίλοφ, Μάρκους Πίπερ και Σον Κέιλι, επόμενη τριάδα. Η Ευγένη όσο πιο σύντομα μπορείς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος, διότι ήθελα να θέσω συγκεκριμένα. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Είστε, πώς να το πω, ε, είναι κοντινή θέση στη δική μας αξιολόγηση. Χαίρομαι που αντιπροσωπεύετε μια νέα χώρα μέλος διότι βλέπω ότι διακρίνεται ξεκάθαρα τη μεγάλη επιρροή που έχει η πολιτική συνοχής στις χώρες της νέες. Όλοι δώσαμε υψηλούς βαθμούς για τα, στα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής μέχρι τώρα. Νομίζουμε ότι είναι επιτυχής. Βεβαίως δεν είναι η ωραία κοιμωμένη. Ε, ε, περιέχει και κάποια προβλήματα. Βλέπουμε σήμερα ότι προσπαθούμε να προσ... γίνεται προσπάθεια να μειωθεί το βάρος της πολιτικής. Η μείωση των πληρωμών κατά ένα δισεκατομμύρια ευρώ είναι κάτι απαράδεκτο. Όχι όσον αφορά μόνο τις οικονομικές συνέπειες, αλλά είναι πολιτικό μήνυμα. Και καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι βλέπουμε και κάποια σημάδια απογοήτευσης, ένα κλίμα απογοήτευσης αρχίζει να επικρατεί. Και ανησυχώ μήπως αυτό το κλίμα οδηγήσει σε κάποια εξαφάνιση της έννοιας της αλληλεγγύης, που σε κάποιους κύκλους ε, γίνεται κακή λέξη η αλληλεγγύη. Γίνεται ύβρις και βλέπουμε την πολιτική συνοχή σαν μια δοκιμή, διότι η έλλειψη αλληλεγγύης θα μπορούσε να επιφέρει ε, μια διαφορετική κατάσταση στην Ένωση στο μέλλον. Και ελπίζω πραγματικά, κύριε Επίτροπε, ότι δεν θέλουμε να έχουμε μεγάλους ιτημένους, αλλά ελπίζω να μην χάσουν τελικά, να μην είναι στους μεγάλους ιτημένους τα νέα κράτη-μέλη. Ο κύριος Πίπερ έχει το λόγο. Ja, vielen Dank. Zunächst eine Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να κάνω μία σύντομη παρατήρηση σε σχέση με το ΑΕΠ. Είναι καθυσιαστικό αυτό το οποίο είπε η Κομισιόν, αλλιώς θα, αλλιώς θα μπορούσαν να επωφεληθούν περισσότερο αυτοί οι οποίοι έχουν εφάνταστη ικανότητα να αλλάζουν τις στατιστικές και να εκμεταλλεύονται τους διάφορους δείκτες. Ένα ερώτημα τώρα για το μηχανισμό επιβολής κυρώσεων. Αντίθετα από άλλους, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένας αυτόματος μηχανισμός ο οποίος ενεργοποιεί αυτές τις κυρώσεις, αλλά όχι στο Ταμείο Συνοχής, αλλά σε, άλλες, ε, σε άλλα κονδύλια. Υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες ήδη στο Ταμείο Συνοχής που δεν τις χρησιμοποιούμε. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιούμε άλλες κυρώσεις. Τώρα, ο, το Ταμείο για την Διάσωση στη ζώνη του ευρώ έχει χρόνο διάρκειας τρία χρόνια. Τι γίνεται μετά και τι σκέφτεστε σε σχέση με την πρόταση που έχει έρθει από την Οικονομική Επιτροπή για μια μέσα σε εισαγωγικά οργανωμένη χρεοκοπία σε κρατικό επίπεδο. Ποια είναι η στάση της Κομισιόν σε σχέση με μια τέτοια δυνατότητα. επόμενος. Α, συγγνώμη, ήμουν σε λάθο θέση, κύριε Δαμίδη. Λέει ο Σκέλη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Υπήρξε πολύ ειλικρινή. Παρουσίασε συνοπτικά την κατάσταση, τη θέση του. Θα προσπαθήσω να είμαι εξίσου σύντομο κι εγώ. Πρώτα απ' όλα, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Χρειαζόμαστε ιδίου πόρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμφωνώ ότι ποτέ δεν θα είμαστε θέση να μιλήσουμε μια φωνή ή να δράσουμε σαν ένα σώμα εάν δεν υπάρξουν κατάλληλα μέσα που θα μας ε, βοηθήσουν να πετύχουμε κάποια μορφή ανεξάρτητης χρηματοδοτήσεως. Ερώτηση. Εξέτασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια μέσα που θα μπορούσαν να σχετικά χρήσιμα. Αποκλείσατε τη φορολόγηση. Τι γίνεται με τα ευρωομόλογα. Διότι πρέπει να πολεμήσουμε κάποια μάχη πάνω σε αυτό. Και πρέπει να ξέρουμε πότε. Αναφέρθηκε μετά στο θέμα μειώσεως των κονδυλίων για τον πολιτισμό. Μπορεί να μας εξηγήσει. Τώρα θα γίνει μείωση. Πόσο. Ποια η άποψή του. Και κάτι ανάλογο και για τη χρηματοδότηση της συνοχής. ΑΕΠ είναι δύσκολο καθόδες θέμα. Η επίμαχο βλέπει κάποια πιθανότητα ότι αν υπάρξουν άλλα στοιχεία, ότι θα ληφθούν υπόψη άλλα στοιχεία πέρα του ΑΕΠ αν θεωρηθούν χρήσιμα. Ο αθλητισμός και ο τουρισμός μετά συμπεριληφθήκαν, δίνονται κάποιες ε, εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της συνθήκης της, Ευρω... της Λισαβόνας. Έχουν, θα υποβληθούν προτάσεις σχετικές. Και ποιες είναι οι οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν και για τον αθλητισμό και για τον τουρισμό. Συμφωνώ επίσης για την εφταετή θητεία, επταετή θητεία. Η θητεία επταετή είναι ιδανική και κρίμα που δεν συμπεριελήφθη στη συνθήκη τη Λισαβόνα και για το Κοινοβούλιο και για τους άλλου φορεί που προτάθηκε. Έλιο Ροκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, λέει ο συνάδελφό ο ο Επίτροπος Ζαχάνε Αάν, δημοσία, πρότεινε κάποια πράγματα αναδόμηση των διαφόρων ευρωπαϊκών ταμείων και νέο στόχο όσον αφορά την αναπτυξιακή πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης προς τις μεγάλες πόλεις, προς τις Μητροπόλεις. Ερώτημα. Πώς θα μεταφραστεί αυτό ε, σε προϋπολογισμό, σε όρους προϋπολογισμού. Στις περιφέρειες στόχου 1 και στόχου 2 Εκεί θα μειωθούν οι πιστώσεις. Στο έγγραφο το σχετικό για τον προπολογισμό είδα ότι για τις πιστώσεις του στόχου 1 προβλέπεται μία μείωση. Μήπως υπάρχει ασυνέπεια εδώ. Να δηλώνει κανείς την ανάγκη να βοηθηθούν οι περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να καλύψουν την καθυστέρησή τους και γι' αυτό δημιουργήθηκαν και τα κριτήρια στόχου 1 και στόχου 2, αυτό από τη μία, και από την άλλη να μειώνονται οι πιστώσεις. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που έχω να σας θέσω, κύριε Επίτροπε. Ο Επίτροπος... Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ναι, εγώ θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Βέβαια, όπως είναι τώρα τα πράγματα, είναι πολύ ευνοϊκή η θέση μου, γιατί μπορώ να επιλέξω πού θα απαντήσω και πού θα δώσω έμφαση. Ο κύριος Κυρίλοφ. Κατανοώ απόλυτα τις ανησυχίες του και τα επιχείρηματά του. Στο τωρινό οικονομικό κλίμα, τι σημαίνουν όλα αυτά. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός αντιμετωπίζεται από πολλούς ως ένας προϋπολογισμός για τους ευρωκράτες και μόνο. Θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια, ένα εγχείρημα δημοσίων σχέσεων και να τονίσουμε ότι αφορά και τους φοιτητές του Εράσμους, τις τοπικές επενδύσεις, τους μη κυβερνητικού ε, φορείς, ε, τη δημιουργία θέσεων απασχόληση σε περιφερειακό επίπεδο, ότι δεν είναι χρήματα για τους ευρωκράτες μονάχα, ότι δίνουν προσθέμενη αξία τα εργαλεία μας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και όχι μονάχα σε εθνικό επίπεδο. Αλλά αυτό δεν είναι μια κοινή θέση. Πολλοί δεν βλέπουν με αυτόν τον τρόπο αυτά τα χρήματα παρά μόνο σαν χρήματα που πηγαίνουν στις Βρυξέλλε. Για το ερώτημα του κύριου Πίπα για τις ε, κυρώσεις. Οι κυρώσει λειτουργούν όταν είναι αυτόματες. <clears throat> ναι, αλλά χρειάζεται κάποιος τζόγο, κάποιο περιθώριο. Και όχι διακριτική ε, διακριτική ανοχή όπως έγινε παραδείγματος το 2004. Αν είμαστε άκαμπτοι, και απάντησα σε αυτό στην κυρία Κρέλ, ότι θα μπορούσαμε να επιδεινώσουμε σοβαρά την θέση ορισμένων χωρών. Αλλά οι κυρώσει θα πρέπει να αφορούν τους υπουργού οικονομικών και όχι τους τελικούς αποδέκτες των κονδύλιων. Αν υπάρχουν κυρώσεις οι οποίες αφορούν όχι μόνο το Ταμείο Συνοχής, αλλά όλες τις, πιστεύω όλες τις όλα τα μεταφερόμενα κονδύλια θα πρέπει να, να αντιμετωπιστούν. Και υπάρχει μια αμφισβήτηση για τα θέματα αυτά, μια διαμάχη στην Κομισιόν, γιατί υπήρχε η δυνατότητα με τους κανονισμούς που είναι ενισχύ να τεθούν κυρώσεις, αλλά δεν τέθηκαν ποτέ κυρώσεις, εκτός από μια περίπτωση στη Βουλγαρία, αλλά και για διαφορετικού λόγου. Χρειάζεται λοιπόν μια πολιτική θέληση για να διαμορφωθούν με τον σωστό τρόπο οι κυρώσει. Αν θα πρέπει να είναι αυτόματοι και άκαμπτη από μία άποψη, αλλά να μην θίγουν περιοχές όπου θα θίξουν τον τελικό αποδέκτη των κονδυλίων αυτό. <clears throat> Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να έχουμε τέτοιους διορθωτικούς μηχανισμούς οι οποίοι θα παίξουν ένα τέτοιο ρόλο σε ό,τι αφορά το Ταμείο Σταθεροποίησης. Αυτό είναι ένα προσωρινό ταμείο για τη ζώνη του ευρώ. Νομίζω ότι αυτή ήταν και η θέση γερμανική στην αρχή ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει ο κίνδυνος να πληρώνει στο διηνεκές και για τους άλλους. Αυτό θα ήταν μια πολύ ευρία ερμηνεία της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Προς το παρόν λοιπόν είναι τριετές το Ταμείο Σταθεροποίησης στη ζώνη του ευρώ και δεν υπάρχει κάποια επίσημη αίτηση να παραταθεί αυτός ο μηχανισμός. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος βασίζεται στην παροχή εγγυήσεων για την δανειοδότηση για τρία χρόνια. Εγώ μπορώ να δεχτώ κάτι τέτοιο αν υπάρξει μια άλλη χώρα πέραν της Ελλάδος η οποία θα ζητήσει χρήματα, αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε μια ανάγκη να παρατείνουμε και πέραν των τριών ετών αυτό το μηχανισμό. Ας ελπίσουμε όμως ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία βρέθηκε σε επιτακτική ανάγκη βοήθειας και κινητοποιήθηκε αυτός ο μηχανισμός. Ακόμα και αν κινητοποιείται ένα τέτοιο μηχανισμός, αυτό δεν σημαίνει ότι θα εμπλακεί αμέσως ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε ένα ειδικό ταμείο για τρία χρόνια και όχι παραπάνω. Κύριε Κέλλη, θέσατε τόσα πολλά ερωτήματα Ίσως θα ήταν πιο εύκολο να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα σε διμερή βάση, καθώς συναντιόμαστε σε διάφορες επιτροπές, για να μπορέσω να διεξέλθω όλα τα ερωτήματά σας. <clears throat> Ξεκινήσατε με το θέμα των ιδιών πόρων. Αυτό είναι τόσο επίμαχο αυτή τη στιγμή, που προτιμώ να μην το θίξω καθόλου. Για να μην με, με γράψουν πάλι οι κύριοι οι τίτλοι των εφημερίδων ότι η Ευρώπη ψάχνει στις τσέπες των πολιτών της για να χρηματοδοτήσει τους ευρωκράτες. Εγώ ελπίζω ότι σε μακροπρόθεσμο επίπεδο θα υπάρξει και κάποια σταθερότητα που να εξασφαλιστεί όχι μόνο επί τη βάση των εθνικών συνεισφορών αλλά και άλλων μορφών φορολογίας. Ο Άντριου Χάμιλτον και οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτών είχαν τονίσει ότι δεν μπορεί να υπάρχει οικονομική διακυβέρνηση αν βασίζεται κανείς μονάχα στην χρηματοδότηση που μεταφέρεται από τα κρατήδια. Αλλά απάντησε ο κύριος Μπράουν ότι την τελευταία φορά που προσπαθήσαμε να έχουμε νέα φορολογία, το αποτέλεσμα ήταν η ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι η απάντηση του Γκόρντον Μπράουν στο επιχείρημα αυτό για το ότι είναι απαραίτητη φορολογία για να εξασφαλίσει την οικονομική διακυβέρνηση. Σας παρακαλώ να είσαστε ε, ανεκτικός γιατί βλέπω να με σπρώχνει, να με πιέζει η Τανούτα. Θέσατε 7 ερωτήματα. Θα τα πούμε προσωπικά, διμερός για να μπορέσω να απαντήσω και στους άλλους ε, ομιλητές, τον κύριο Ορό. Αυτή τη στιγμή είναι υποσυζήτηση ένας μηχανισμός που αφορά τις αστικές συγκεντρώσεις. Φυσικά δεν μπορεί να είναι ο κύριος στόχος μας. <clears throat> Γιατί οι αστικοί αυτοί οι χώροι που περιλαμβάνουν τη Βαρσοβία έχουν πολλά προβλήματα. Δεν μπορώ να σας πω σήμερα πώς θα διαρθρωθεί αυτή η χρηματοδότηση, αλλά υπάρχει πρόβλεψη στην πολιτική συνοχή με πέκυνα το 2013 να ληφθούν υπόψη οι, αστικοί, ε, οι αστικές συγκεντρώσεις. Θα έρθει και από εμά ένα έγγραφο στρατηγικής για την συνοχή. Αυτό το έγγραφο που περιλαμβάνει και τους αστικούς χώρους θα δημοσιευτεί το Νοέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου ίσως, και αυτό το στρατηγικό έγγραφο για τη συνοχή μετά από το 2013 θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια λύση, η οποία είναι τώρα υπό τεχνική επεξεργασία για τις μεγάλες πόλεις. Ο Ιωάννης Χάντς, Χάνες νομίζω ότι υποστηρίζει κάτι τέτοιο και ήταν η δική του πρόταση εφόσον έρχεται από μια μεγάλη πολιτική Βιέννη να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά φυσικά δεν είναι ο πρώτος μας, πρωταρχικός μας στόχος. Ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα τον κύριο Κέλλη που δεν μπορώ να απαντήσω στα ερωτήματά του. Απλώς σας λέω ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα των ιδιών πόρων. Έχουμε ακόμη τέσσερις ομιλητές. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα σύντομοι. Ο κύριος Φανίστερ Ρόι συντονιστής για την ομάδα του ΕΛΚ στην Επιτροπή Ενέργειας. Λοιπόν. Και έχουμε και άλλου τρει ομιλητέ. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε πολύ σύντομοι γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο σημείο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να προβλέψουμε και άλλη συνάντηση με τον κύριο Επίτροπο. Διότι Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολλά αυτά που έχουμε να συζητήσουμε. Τώρα μιλάμε για την περίοδο 2014-2020 ήδη. Την τελευταία φορά είχαμε συζητήσει επί πολύ μεγάλο διάστημα για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και είχαμε και δυσκολίες υλοποίησης από των υστέρων. Το ίδιο λοιπόν μπορεί να συμβεί και με την επόμενη περίοδο των δημοσιονομικών προοπτικών. Είναι λοιπόν τα πάντα θέμα προγραμματισμού. Μιλάμε για την πολιτική συνοχής προφανώς, αλλά θα πρέπει επίσης να διδαχθούμε και από τα σφάλματα του παρελθόντος. Υπήρχε μια εσωτερική ομάδα εργασία η οποία ασχολήθηκε επισταμένα με το όλο ζήτημα των δημοσιονομικών προοπτικών. Τώρα μα ενδιαφέρει Πώς λοιπόν θα οργανωθούμε από πλευράς Κοινοβουλίου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να έχουμε μια εδαφική πολιτική, πολιτική συνοχής επιτυχημένη, εάν δεν συμπεριληφθούν όλες οι περιοχές της Ευρώπης. Άρα μιλάμε για επενδύσεις προς όλες τις περιοχές. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης κάλυψη. Και βεβαίω αυτό δεν πρέπει να το δει κανεί αρνητικά. Σίγουρα ο καθένα θέλει την ανάπτυξη να την ε, ενθαρρύνει προ όφελό του, αλλά όλοι θέλουν και να ωφεληθούν από τι ε, πολιτικέ μα. Αυτό σαφώ δεν το ξεχνάμε. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε στι συζητήσει με το θέμα. Είναι λοιπόν νομίζω σημαντικό να συνεχίσουμε να δούμε πώς θα έχουμε μια ορθή προσέγγιση από πλευράς Κοινοβουλίου. Για τα διάφορα προγράμματα και τη χρηματοδότησή του, λοιπόν. Εδώ μιλάμε για μεγάλε υποδομέ, υποδομέ διασυνοριακές, διακρατικέ, αλλά πολλέ φορέ λείπουν τα κονδύλια. Πώ θα συμπληρώσουμε, λοιπόν, τα ελλείμματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο κύριος Σαμπαρόζο το ανέφερε στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης. Δεν θα επιμείνει να περιπτέρω, απλώς περισσότερα κονδύλια για τα προγράμματα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και να θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα και μόνο. Αλλά καταρχήν θέλω να κάνω μια παρατήρηση για τις κυρώσεις. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει νόημα, όπως είπε και ο κύριος Στρόιλερ, να χρησιμοποιούνται τα διαρθρωτικά ταμεία για να αντιμετωπιστούν μακροοικονομικοί στόχοι. Το ερώτημά μου είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με τη χρονική διάρκεια. η Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών έχει ενιαία άποψη. Θεωρεί ότι πέντε χρόνια για τα διαφορετικά ταμεία ως περίοδος προγραμματισμού δεν είναι δυνατή, δεν είναι εφικτή ούτε για την προετοιμασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε για τις περιοχές που είναι οι αποδέκτριες. Δεν μπορώ να φανταστώ λοιπόν να υπάρξει μια τέτοια ρύθμιση για πέντε χρόνια μονάχα. Και είμαι αρκετά χρόνια σε αυτό το κοινοβούλιο και είχε υπάρξει πενταετής περίοδος προϋπολογισμού στη δεκαετία των 1990 και καταργήθηκε γιατί δεν έχει νόημα. Επίσης, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, υπάρχουν μια σειρά από καινοτομίε στο να προσδιορίζονται συγκεκριμένα χρήματα για ορισμένες ενέργειες. Η Κομισιόν δεν φαίνεται να το υποστηρίζει αυτό το πράγμα. Ποια είναι η άποψή σας τώρα για αυτό το λεγόμενο ring financing, Δηλαδή, να υπάρχουν χρήματα τα οποία προσδιορίζονται για συγκεκριμένους στόχους. Όταν πρόκειται παραγωγός χάρη για τις ανανεώσιμες ενέργειες, για την εξυγίανση των κτηρίων, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το δεχτεί η Κομισιόν ή είναι κάτι στο οποίο αντιτίθεστε από, απόλυτα. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Είναι γνωστό ότι εσείς θέλετε να ενοποιηθούν οι, μηχανισμοί δημοσιονομικού ελέγχου και αν πάρουμε σαν παράδειγμα τα, πο, τα ποσά που δίνονται για τη γεωργία. Εγώ πιστεύω ότι αυτά δεν έχουν λειτουργήσει τα θέματα δημοσιονομικού ελέγχου, ιδίως για τα μικρά προγράμματα και ίσως θα έπρεπε να έχετε και μία έκθεση ε, αντικτύπου για να δείτε αν μπορείτε να διαχειρίσετε αυτά τα προγράμματα ή πρέπει να υπάρχει μια πιο κεντρική διαχείριση. Ο Τζιβλάσα και μετά ο Ρικάρντο. Ευχαριστώ αγαπητέ Επίτροπε και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που μας δίδεται δυνατό της ε, διεξαγωγής της συζητήσεως και ότι θεωρείται την πολιτική συνοχή σαν κάτι σημαντικό. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αν θέλουμε οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να βρούμε πόρους και αν 70 ή 80% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ προέρχεται από τις μεγάλες πόλεις και τις αστικές περιοχές, θα πρέπει να ρωτήσουμε αυτές τις μεγάλες πόλεις κατά πόσο χρειάζονται βοήθεια. Εάν έχουν προβλήματα. Πώς θα δράσουμε λοιπόν σαν εταίροι αυτών των πόλεων στο μέλλον. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτή η μεγάλη δήμη επίσης θα βοηθηθούν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα όσον αφορά την εφαρμογή της εξοικονόμησης ενέργειας, ασφαλή φοδιασμό ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας κλπ. Αν θέλουμε να κάνουμε περικοπές, έχουμε τους μεγάλους δήμους και τις πόλεις που μπορούν να κάνουν οικονομίες εύκολα αν χρησιμοποιήσουν περιβολαντικά φιλικές μεταφορές, ε, φωτισμό, ε, πράσινα κτίρια. Ερώτηση, θα βοηθήσουμε τις πόλεις στο μέλλον. Δίνοντας περισσότερους πόρους να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Τελευταίο ερώτημα που συνεχίζει το ερώτημα της κυρία Μανέσκου που έθεσε κάτι πολύ σημαντικό για κάποια κατάρτιση της τοπικής αυτοδίκησης των ανθρώπων που ζουν στους Δήμους και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είχαμε συζητήσει ένα ενδεχόμενο πρόγραμμα έρασμος για τους ε, υπαλλήλους των Δήμων. Ε, ποια είναι η απόψή σας που στηρίζετε τέτοιο μέτρο. Επόμενος. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Πετροπέ, που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας. Πρώτα απ' όλα, Νομίζω ότι καθίσταται σαφέ ότι η Επιτροπή, η μας έχει αρκετά ενιαία στάσεις ό,τι αφορά την, ε, τον προπολογισμό. Αύριο θα ψηφίσουμε για ένα προφορικό ερώτημα που ελπίζουμε θα μπορέσουμε να υποβάλουμε στην, επόλη, στην επόμενη μήνυ ολομέλεια και στην τρίτη παράγραφο του ερωτήματο αυτού φροντίζουμε να γίνει σαφέ ότι το να υπάρχει εύρωστη περιφερειακή πολιτική και πολιτική συνοχή μέσω στη χρηματοδότηση για την Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό, εάν θέλουμε να πετύχουμε πραγματική εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι και το όλο θέμα. Και εσεί στα σχόλιά σα ε, είπατε ότι προσυπογράφετε πλήρω σε μια τέτοια προσέγγιση. Θα ήθελα να σχολιάσω ένα-δυο από τα σημεία που εσείς αναπτύξατε, δεδομένου του κλίματος απεσιοδοξίας που φαίνεται να κυριαρχεί στην Ευρώπη, όπως είπατε. Υπάρχει λοιπόν πολύ σκεπτικισμός, ακριβώς γιατί φαίνεται η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να πηγαίνει για κά... κατά την άποψη κάποιων στις τσέπες των ε, ευρωκρατών. Αυτό βεβαίως ε, φαίνεται να υπονομεύει και τον σχεδιασμό του προπολογισμού. Δεν θέλω βεβαίω να συνοψίσω τα όσα είπατε με αυτέ τι δύο κουβέντε, όμω αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην εξαιρετική σα παρουσίαση δεν θέλετε να μιλήσετε για του ιδίου πόρου. Εντάξει, αλλά στο μέλλον μπορεί ήδη αυτοί που όλοι να συσχετιστούν με την ε, πολιτική συνοχή, με την παραγωγική πολιτική. Θα μπορούν όλοι οι πολίτες της Ευρώπης να παρακολουθούν πώς οι οι πόροι διοχετεύονται στα προγράμματα αυτά που ευεργετούν, ωφελούν ακριβώς τους ίδιους τους πολίτες και μάλιστα άμεσα. Και κάτι για τις ε, μεγάλες, τις ευρύτερες περιφέρειες Πιστεύετε ότι στο μέλλον θα έχουν συγκεκριμένα κονδύλια που θα τους αποδίδονται οι περιοχές αυτές. Oh, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Κύριε Βανίστερ Για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην περιφερειακή πολιτική έχω την ίδια θέση με σας. Αλλά όπως ακούσαμε και από την κυρία Μανέσκου, Είπαμε, είπε και εκείνη ότι πρέπει να υπάρχει διάδοση των καλύτερων προτύπων ε, για τον προγραμματισμό, για τον έλεγχο, κατάρτιση λοιπόν των ε, λειτουργών της των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτό ιδιαίτερος για την ε, λεγόμενη προανατολική Ευρώπη. Είναι σημαντικό, σημαντικό να υπάρχει μια σωστή νοοτροπία για τους ελέγχους για την δαπάνη των ε, κονδυλίων. Χρειάζεται αυτό για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και για τα ευρωμόλογα που ανέφερε και ο κύριος Μπαρόζο στην ομιλία του για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωση. Εδώ μιλήσαμε αρχικά για τις χώρες που έχουν προβλήματα ε, στην περίπτωση της λύσης Ιούγκερ. αλλά το θέμα είναι πώς θα επιτραπούν, επιτραπεί ο δανεισμός σε χώρες που χρειάζονται ακριβώς τέτοιου είδου στήριξη. Και το θέμα είναι τι θα γίνει και με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Πέραν των μεταφορών και για την ενέργεια. Εκεί είδαμε πώς μπορεί να επεκταθεί ο προπολογισμό. Το αποτέλεσμα για τον προπολογισμό όμω δεν αλλάζει σοβαρά. Δηλαδή, αν για τον ισολογισμό υπάρχουν συνέπειες από τον μηχανισμό σταθεροποίησης και ένα κουτί εργαλείων με κυρώσεις, ε, και πάλι αν ε, πολιθούν ευρωομόλογα, η Επιτροπή δεν θα λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, θα είναι κάτι παράπλευρο αυτό που θα συμβεί στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Εκεί η διαμεσολαβητής θα είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ο Ευρωπαϊκός Προεπολογισμός λοιπόν ε, σαφώς θα επηρεαστεί όσο καλή και αν, είναι αυτή η ιδέα, αυτή η σύλληψη των ευρωομολόγων. Πάντως ε, θα ήταν ακριβώς το ίδιο το αποτέλεσμα με, τις, ε, με το δανεισμό του τύπου Juncker. Τώρα, για τη μακροσκελή περίοδο προγραμματισμού και για το αν θα έπρεπε να είναι συντομότερη. Ναι. Είμαστε στο τέταρτο έτος της τρέχουσας ε, περίοδου δημοσιονομικών προοπτικών. Το 2010 ήταν το τέταρτο έτος. Και μόνο τώρα φτάσαμε μια σωστή ταχύτητα στην πολιτική συνοχή. Στα τρία χρόνια ήταν σχεδόν η αρχή, το ζέσταμα. Ο τέταρτος χρόνο, στο τέταρτο έτος, είναι σχεδόν στο τέλος της πενταετούς περίοδου. Και η πρακτική μας εμπειρία τι μας λέει, ότι δεν ήταν κακή η ανακάλυψη η επταετία για τον προγραμματισμό και για την ε, υλοποίηση των υποσχέσεων που είχαν δοθεί στις περιφέρειες της Ευρώπης. Δεν θυμάμαι να υπήρξαν δυσκολίες με την έρευνα για να απαντήσω και σε αυτό το ερώτημα. Τώρα, τι προβλήματα προβλέπονται μελλοντικά από το 2013 και μετά για την έρευνα και για τα ευρεία κλίμακα προγράμματα. Το ίντερ είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και η χρηματοδότησή, μου, χρηματοδότησή του για το 2012-2013. Τέτοιου είδου δαπάνε, τέτοιου είδους κονδύλια που γοργά ε, αυξάνοντας προς το κόστος, διότι το ΙΤΕΡ προβλεπόταν για 5 δις ευρώ στη φάση οικοδόμησης και τώρα έχει φτάσει τα 15. Οι επιστήμονές μας αρέσκονται στο να αυξάνουν και να πληθαίνουν το κόστος. Αυτό λοιπόν από άποψη προγραμματισμού του προπολογισμού είναι σπαζοκεφαλιά. Δεν μιλάμε για 1% ή 2% αύξηση. Από τα 5 στα 15 δις έχουμε φτάσει. Πάντω δεν θα υπάρξουν δυσκολίε με τα μικρή εμβέλεια προγράμματα από το 2013 και μετά. Νομίζω ότι θα παραμείνουν όσοι είχαν. Και για το μοντέλο άκρα θα πρέπει και στις εθνικές δηλώσεις να δούμε τι αποτελέσματα τύπου σχέσει μπορούν να δοθούν που να είναι εφικτέ. Ε, δηλαδή η ομοσπονδιακή οικοδόμηση τη Γερμανία, σε κρατήδια, σε Λάντερ, είναι ένα παράδειγμα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη γεωργία, με τι εκταμιεύσει, με του οργανισμού που χειρίζονται τα κονδύλια τοπικά. Αυτό όμω είναι μια φιλοδοξία πολύ ψηλή και ίσως να τεθεί το θέμα στην ε, μετά από τριετία αναθεώρηση. Ο κύριος Βλάση ξέρω ότι είναι εισηγητής για την αναπτύξη της υπαίθρου και δυστυχώ ε, η παρέμβασή σας ήρθε πολύ καθυστερημένα στην όλη μα συζήτηση από άποψη χρόνου. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω λοιπόν κι άλλο Παρατείνοντα την αναμονή σας και μακρηγορώντα για να σα απαντήσω. Πάντω αν θέλουμε από τα εξοικονόμηση ενέργειας στην Ευρώπη, πέραν των ανανεώσιμων πηγών, ο βασικός τομέας που πρέπει να επικεντρωθούμε είναι η στέγαση, τα κτίρια. Εκεί υπάρχει πραγματική δαπάνη, υπάρχει πραγματική κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη. Και για να ολοκληρώσω με τον κύριο Κόρτες Λάστα, δεν συζητάμε μόνο για τους ιδίου πόρους, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι τα χρήματα που πήγαν από μια συγκεκριμένη πηγή δαπανήθηκαν για τον πολύ συγκεκριμένο στόχο για τον οποίο προορίζονταν. Η λογική λοιπόν του προπολογισμού είναι αυτή, ότι πρέπει να υπάρχει μια τέτοια εξέταση των κονδυλίων. Όμως αυτό προκαλεί και προβλήματα σε περιοχές που έχουν ιδίους αλλά έχουν και συγκεκριμένο στόχο, δαπάνη που τους αποδίδεται. Υπάρχουν λοιπόν περιοχές όπου ήδη έχει σημειωθεί, έχει αποσταλεί κονδύλι της Επιτροπής, αλλά υπάρχουν και έσοδα από πώληση δικαιωμάτων ε, εκπομπής διοξυδίου του άνθρακα. Φαίνεται λοιπόν ότι ακόμη υπάρχουν ατέλειες και βλέπετε ότι είναι πολλά αυτά που απομένουμε να κάνουμε για να καλύψουμε τις ελλείψεις μας. Ε, με συγχωρείτε για τις βιασμένες κάπως απαντήσεις μου στις ερωτήσεις σας. Ξέχασα ίσως την δεύτερη, αλλά νομίζω θα ήθελα να επιδείξω την ίδια επιμέλεια που έδειξε ο κύριος Κέλλη Νομίζω ότι ήταν ο πιο ταχύ από του ομιλητέ σας. Κατάφερα να απαντήσω το ένα από τα έξι ερωτήματα του μόλι. Ευχαριστώ Επίτροπε εκ μέρου μα σα ευχαριστούμε για την πραγματικά ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων για ένα θέμα που είναι τεράστια πρόκληση για όλου μα και στο Κοινοβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτιμώ την ετοιμότητά σα να αναφερθείτε στι μεγάλε προκλήσει τη πολιτική συνοχή και να επισέθετε σε πολλέ λεπτομέρειε όσον αφορά την πολιτική συνοχή και ελπίζουμε ότι αυτό σας επιτρέπει να καταλάβετε και να ανταποκριθείτε καλύτερα, ελπίζουμε, στις ανησυχίες μας. Αναλάβατε την υποχρέωση αντι του Σον Κέλλη να έχετε ένα πρόγευμα εργασίας για να απαντήσει ερωτήσεις του, αλλά με τα χαράς να σας φιλοξενήσουμε εκ νέου στο εγγύς μέλλον για να συνεχιστούν οι συζητήσεις όσον αφορά το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε. Που πλησιάζει τις θέσεις μας όσον αφορά τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής. Θεωρούμε επίσης ότι είστε φίλος της πολιτικής συνοχής, αυτό σας χαρακτηρίζει και νομίζω ότι θα είσαστε ανοιχτός για να απαντήσετε σε ερωτήσεις μας στο μέλλον σας ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να μείνετε, αλλά θα καταλάβουμε επίσης αν υποχρεωθείτε να αποχωρήσετε. Uh, Και τώρα, χωρίς διάλειμμα, προχωράμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Είναι μήνυα ακρόαση που σχετίζεται με την, έκθεση πρωτοβουλίας του Ότζι Βλάσακ που προετοιμάζεται αυτή η έκθεση. Δεν έχουμε κάποιο έγγραφο εργασίας. Έχουμε δύο έξοχους εμπειρογνώμονες μαζί μας, ότζι για να συντομεύουμε, θα το λόγο, για να μας παρουσιάσει τους φιλοξενούμενούς μας και να κάνεις μια εισαγωγή στην συζήτηση. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στην αρχή επιτρέψτε μου να παρουσιάσω μια εισαγωγή στο κείμενο, το οποίο σας έχω διανύμει. Πρόκειται περί μιας πρώτης συζητήσεως για τη μελλοντική έκθεσή μας, με θέμα τη μελλοντική έκθεσή μας, για το Ευρωπαϊκό Αστικό Περιβάλλον, πρόγραμμα για το Ευρωπαϊκό Αστικό Περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή. Είναι κάτι που θα συζητηθεί. Και σας με αυτό το έγγραφο κάποια από αυτά τα θέματα και ίσως να αποτελούν πρόκληση. Θα ήθελα να μελετήσετε το έγγραφο που σας μοίρασα όμως και αν τυχόν έχετε κάποιες ιδέες, κάποιες προτεραιότητες, ελεύθερα ας έρθετε σε επαφή μαζί μου μέσω email ή πρόσωπο με πρόσωπο. Πιστεύω ότι τα βασικά θέματα προς συζήτηση θα πρέπει να είναι τα εξής. Πρώτον, αστικές προκλήσεις, προκλήσεις της πόλης. Όλοι καταλαβαίνουν ότι στην Ευρώπη έχουμε πληθυσμό περίπου 500 εκατομμύρια. Και όπως προανέφερα, σχεδόν 80% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγεται στις πόλεις και τις αστικές περιοχές. 80% των κατοίκων της Ευρώπης κατοικούν σε αστικές περιοχές και σε πόλεις. Άρα οι πόλεις μας χρήζουν προσοχής. Και γι' αυτό θα πρέπει να εντοπίσουμε τα βασικά θέματα προς συζήτηση. Ποιες είναι οι ανάγκες των πόλεων. Τι προκλήσεις αντιμετωπίζονται από τις πόλεις. Τι προτεραιότητες έχουν οι πόλεις. Και αυτές οι προτεραιότητες ταιριάζουν με τις προτεραιότητες που περιέχονται η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το 2020. Τι μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έχουμε τα κατάλληλα μέσα. Ή θα πρέπει να αντικατασταθούν από κάποια μέσα που θα εξυπηρετούν καλύτερα τους σκοπούς μας. Επόμενο ζήτημα είναι της αναθέσεως κάποιων ευθυνών, εκχωρήσεως ευθυνών. Μπορούν να εκχωρηθούν στους Δήμους οι ευθύνες για τη διαχείριση των πόλεων. Στη μήνυα ακρόασή μας λοιπόν θα μπορέσετε να ακούσετε σχετικά παραδείγματα που θα δείχνουν πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι που διατίθεται από πόλεις και ποιο ποσοστό των πόρων θα πρέπει να χορηγείται μέσω χορηγιών και ποιο ποσοστό θα πρέπει να χειρίζονται άλλα οικονομικά μέσα. Θα πρέπει και τις συνεργασίες να τις συζητήσουμε σε σχέση με το θέμα αυτό. Το ερώτημα που απευθύνθηκε προς τον Επίτροπο αφορούσε ακριβώς αυτό. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τις μεγάλες πόλεις και τις αστικές περιοχές να μας πούν γιατί χρειάζονται τα χρήματα. Πρέπει να ξέρουμε τι ανάγκες θα αντιμετωπιστούν. Θα πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσουμε κατά πόσο η ε, χώριση δικαιοδοσιών είναι, θα είναι κάτι υποχρεωτικό ή θα εφαρμόζεται θελοντικά. Μετά, χρηματοδότηση. Άλλο θέμα αυτό. Πάντα τα χρήματα έχουν προτεραιότητα και κάποιο ποσοστό των πόρων δεν χρησιμοποιείται πλήρως. Υπάρχουν κάποια μέσα που δεν χρησιμοποιούνται όσο θα ήταν δυνατόν, όπως τα μέσα Jessica. τι μέθοδο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ποια εμπόδια υπάρχουν, ποια εμπόδια σταμάτησαν τις, τη σωστή εφαρμογή αυτών των μέσων, τι μπορεί να γίνει στο μέλλον για να χρησιμοποιηθούν καλύτερα οι πόροι με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Υπάρχουν άλλες δυνατότητες. Κάτι μεταξύ χωριών και του μέσου. Τζέσικα, μήπως μπορούμε να εφεύρουμε κάτι καινούριο, κάποια κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τις πόλεις να ζητήσουν τη χρήση αυτών των μέσων. Τελικό σχόλιο όσον αφορά τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Ήδη έχουμε καταλήξει σε κάποια συμφωνία. Όλοι θεωρούμε ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση, ο ολοκληρωμένο σχεδιασμό είναι προαπαιτούμενο. Έχουμε εισαγάγει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό όσον αφορά την αστική ανάπτυξη και θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε σε ποιο βαθμό αυτή η προσέγγιση υπήρξε επιτυχής στην εφαρμογή της. Και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός πιστεύω θα γίνεται όλο και πιο σημαντικό στο μέλλον. Όμως, Απ' την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει να αποκεντρώνουμε υπερβολικά τη διάθεση των πόρων, να μην έχουμε υπερβολικό κατακαιρματισμό. Αυτά εν είδη εισαγωγή για το θέμα μας. Να σας παρουσιάσω τους δύο φιλοξενούμενους μας που είχαν την καλοσύνη να δεχθούν την πρόσκλησή μας σε αυτή τη μήνυα κρόση, τον κύριο Ρουτ Βαν Ράγκ, διαχειριστής προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και είναι διαχειριστής, διευθυντής προγραμματισμού επίσης για την ε, ανάπτυξη των περιοχών. Είναι ένα πρόγραμμα που δρομολογήθηκε στην Ολλανδία, το οποίο χειρίζεται, που συναθρίζει τις μεγαλύτερες πόλεις, την Ουτρέχτη, τη Χάγη και το Ρότερνταμ, και οι πόλεις αυτές μέσω του φορέα διαχείρισης των προγραμμάτων χειρίζονται πόρους, χρησιμοποιούν πόρους και ο κύριος Ρότβαν Ραγκ θα μας πει ποιες είναι οι εμπειρίες τους όσον αφορά την χρήση αυτών των πόρων. Ο Τζέρι ο κύριος Τζέρι Μαρίγκεν είναι ο δεύτερος φιλοξενούμενος που είναι επικεφαλής της αποστολής της Βορείου ε, Ιρλανδίας στις Βρυξέλλες είχε υψηλές θέσεις στην κυβέρνηση, στις, μάλλον στη διοίκηση της Βορείου Ιρλανδίας και έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Αμέσως λοιπόν θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρουντ Βον Λάγκ για να κάνει την παρουσίασή του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έχω, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την ευκαιρία που έχουμε να παρουσιάσουμε τις εμπειρίες μας και σας ευχαριστώ φυσικά για την πρόσκληση που μας απευθύνετε. Θέλω να σταθώ σε κάποιες από τις ε, εμπειρίες που είχαμε σε αυτή την προγραμματική περίοδο και μετά ίσως μπορούμε να κάνουμε και κάποια συζήτηση για το πώς ε, φαίνονται οι προοπτικές για το μέλλον. Το πρόγραμμά μας είναι οι ευκαιρίες για την Δύση, όπως αναφέρεται. Είναι ένα σύντομο πρόγραμμα σύντομο σε ιστορία έχει να κάνει με τις εμπειρίες των πόλεων της ε, Ολλανδίας με το πρόγραμμα Urban μέχρι το 2006 και στα πλαίσια του διαστήματος προγραμματισμού 2000-2006 είχαμε ένα πρόγραμμα City και στη συνέχεια έπρεπε να δώσουμε μια νέα λύση για την ε, προσέγγιση μας για το πώς μπορούν να ενταχθούν καλύτερα οι πόλεις σε αυτό το σύστημα. Θέλαμε λοιπόν να κρατήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές από το πρόγραμμα Urban και από το ειδικό πρόγραμμα για τις πόλεις, το City, για να τα ενσωματώσουμε σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα. Στην ε, Ολλανδία έχουμε τέσσερις περιοχές για προγράμματα και μόνο στο δυτικό μέρος της Ολλανδίας είναι διαφορετικά τα πράγματα γιατί στο παρελθόν δεν υπήρχε κανένα πρόγραμμα γιατί οι επαρχίες της νότιας και δυτικής Ολλανδίας δεν, δεν ήταν επιλέξιμες για χρηματοδότηση του στόχου 2. Είναι η πρώτη φορά που η Δυτική Ολλανδία παίρνει τέτοια χρηματοδότηση. Λόγω αυτής της κοινή προσέγγισης δεν έχουμε χωριστά προγράμματα city ή περιφερειακού χαρακτήρα. Όλα αυτά πρέπει να ενσωματωθούν στα γενικά προγράμματα που αφορούν διάφορα τμήματα της χώρας μας. Βλέπετε τώρα την περιοχή στο δυτικό μέρος της Ολλανδίας που ισχύει το πρόγραμμά μας, η περιοχή της Ουτρέχτη, ε, Ρότερνταμ, Χάγης και Άμστερνταμ. Καλύπτονται οι τέσσερις λοιπόν μεγάλοι ε, αστικοί ε, συνοικισμοί, μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις στην Ολλανδία. Τώρα, πώς έγινε δυνατόν να λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να ξέρετε ιδιαίτερα την κατάσταση της Δυτικής Ολλανδίας, στη λεγόμενη περιοχή Randstad, όπου είναι δεσπόζουσα η θέση των μεγάλων τεσσάρων πόλεων. Δεν υπήρξε όμως μια δημοκρατική ε, διοικητική οντότητα στο επίπεδο της Ρανστατ. Ε, Μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο πόλεων. Και είπε επίση η Ολλανδία ότι θέλουμε ένα ενιαίο πρόγραμμα για όλη τη δυτική Ολλανδία. Βρήκαν από τους κανονισμούς ότι υπήρχε δυνατότητα για ε, περαιτέρω εκχώρηση, για εκ νέου εγχώρηση αρμοδιοτήτων και υπήρχε δυνατότητα να υπάρχει μια αντιμετώπιση τέτοια για τη Δυτική Ολλανδία που θα μπορούσε να είναι πιο αποφελής από αυτές του παρελθόντος. Είπανε τουλάχιστον για τη Δυτική Ολλανδία θα πρέπει να υπάρχει μονάχα ένα πρόγραμμα περιφερειακού ταμείου και τίποτα περισσότερο. Ξεκίνησε στη συνέχεια διαπραγμάτευση μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών και χρειάστηκαν περίπου δύο χρόνια για να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση για ένα κοινό λειτουργικό πρόγραμμα. Χρειάστηκε να γίνει η ανάλυση των στόχων, των στρατηγικών, των δυνατοτήτων χρηματοδότησης, της οργανωτικής δομής και το θέμα της οργανωτικής δομής, το οποίο ήταν καινο, Φανές ουσιαστικά, ήταν αυτό το οποίο απέσπασε την περισσότερη προσοχή και καταδαπάνησε τον περισσότερο χρόνο. Ποιος λοιπόν θα πρέπει να είναι αρμόδιος για τι θέμα. Βλέπουμε τώρα τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν. Το επόμενο μάλλον, ε, η επόμενη μάλλον διαφάνεια. Καταρχήν δεν υπήρχε η συνήθεια της συνεργασίας σε ένα κοινό πρόγραμμα και αυτό δεν είναι μονάχα στη δική μας ε, περίπτωση. Πολλοί έχουν τέτοια προβλήματα. Οι τέσσερις πόλεις είχαν η κάθε μία μια ισχυρη θέση η στην επαρχία της και υπήρχαν αντιπαραθέσεις όπως μπορεί κανείς να περιμένει, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικοί τρόποι χάραξης πολιτικών ε, κατευθύνσεων. Όλα αυτά είχαν επιρροή στις αρχικές διαπραγματεύσεις, διαφορετικές μεθοδολογίες, διαφορετικές αρμοδιότητες επίσης. Και τέλος, στη συνέχεια των διαπραγματεύσεων τα πράγματα έγιναν πιο απτά και συγκεκριμένα ποιος πληρώνει αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, ποιος φταίει, αν πρέπει κανεί να είναι πιστό στο αφεντικό του μέσα στα πλαίσια συνεργασίας ή πιστό στο συνολικό πρόγραμμα. Οι περισσότεροι από τους φόβους μας τελικά δεν έγιναν πραγματικότητα. Αυτά που φοβόμασταν πριν από 3-4 χρόνια και μας εμπόδισαν να κοιμόμαστε δεν έγιναν πραγματικότητα. Λύσαμε πάρα πολλά προβλήματα. Πώς έγινε αυτή η επίλυση των προβλημάτων. Η βασική αρχή ήταν ότι πρέπει να συμφωνήσουμε. Και καταλήξαμε να έχουμε μνημόνια κατανόησης από όλους τους εμπλεκόμενους που υπεγράφησαν από τους δημάρχους των μεγάλων πόλεων και κατανεμήθηκαν αρμοδιότητες, τρόποι διαιτησίας, δημιουργήθηκαν Επιλήθηκαν διαφορές κτλ. Υπήρξαν δεσμεύσεις σε επίπεδο προϋπολογισμού και κονδυλίων. Η προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί από κάθε περιοχή κτλ. ώστε να έχουμε τη σωστή συγχρηματοδότηση από τους οκτώ δημοσίους φορείς οι οποίοι έπρεπε να εμπλακούν σε αυτό το πρόγραμμα. Έρχομαι τώρα στα ενδιάμεσα, στους ενδιάμεσους φορείς και το πώς λειτουργούν. Να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι γυρίσατε προς τα πίσω τώρα στις διαφάνειες. Α, εδώ είναι το επόμενο. Πολύ ωραία. Οι συμφωνίες για τις τρεις πόλεις υπογράφονται από τους, τους δημάρχους και αφορούν ακριβώς τις δεσμεύσεις και την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων για τις ε, περαιτέρω εκχωρήσεις για τις αστικές περιοχές και μέσα στα πλαίσια της εργαλειοθήκης που επιτρέπει ο κατάλληλος, ο αρμόδιος κανονισμός. Έχουμε λοιπόν χωριστές ευκαιρίες για κάθε πόλη και υπήρξε ένα συνολικό ποσό χρηματοδότησης χορήγησης που δόθηκε και οι εμπλεκόμενες πόλεις συμφωνήσανε στις ε, προϋποθέσεις για χρηματοδότηση και πώς θα αντιμετωπιστούν ε, ατασταλίες ή αντιρρήσεις, πληρωμές κτλ. Υπήρξε λοιπόν μια συμφωνία που κάλυπτε όλους και μετά ειδικέ συμφωνίες για κάθε πόλη και για τις επιμέρους εκχώρησης. Στην επόμενη διαφάνεια η διαχειριστική αρχή είχαμε τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Ρότερνταμ που είχαν την επίσημη ευθύνη διαχείρισης επειδή ήταν ένα πρόγραμμα που εκπονήθηκε από τις ίδιες πόλεις, τελικά επιλέγει το Δημοτικό Συμβούλιο με το Δήμαρχο μιας από τις τέσσερις πόλεις και ενεκρίθη αυτό και από τον Υπουργό Οικονομικών Θεμάτων της ε, Ολλανδίας να έχουν την ευθύνη της εφαρμογής του προγράμματος αυτού για τη Δυτική Ολλανδία. Το Ρότερνταμ είναι η μόνη πόλη μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, δεν είναι περιοχή, είναι η μόνη πόλη που, έχει την, ε, που μπορεί να είναι διαχειριστική αρχή στην Ευρώπη, αλλά οι άλλες τρεις πόλεις πήραν μια εκχώρηση αρμοδιοτήτων ως ενδιάμεση φορείς. και έχουν το χαρακτήρα επομένω ενδιάμεσου φορέα στα πλαίσια αυτής της ενέργεια. Ε, οι ενδιάμεσοι φορείς και αυτοί έχουν τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι προγραμματική αρχή, Επομένω, έχει την ευθύνη για το πρόγραμμα στη δική του πόλη, βάσει της Συμφωνίας δέσμευση και Εφαρμογής που έχει γίνει με τι υπόλοιπε πόλεις. Αντιμετωπίζουν λοιπόν τα συστήματα ελέγχου, τις πιθανές ατασταλίες, τα προβλήματα εφαρμογής στην περιοχή τους. Όπως προβλέπετε από τον κανονισμό λοιπόν, εκχωρούνται οι αρμοδιότητες για τα θέματα αυτά στους ενδιάμεσους φορείς. Η καθημερινή συνεργασία τώρα έχουμε μια, ένα γραφείο διαχειριστικής αρχής που είναι πολύ μικρό με πέντε άτομα μονάχα που συντονίζουν το, συνολικό πρόγραμμα. Υπάρχουν πέντε εκτελεστικά γραφεία προγράμματος, τέσσερα στις τέσσερις πόλεις και ένα πέμπτο για την περιφερειακή πτυχή που αφορά την Ήπεθρο περισσότερο. Τέσσερα σημεία υποστήριξη σε επίπεδο επαρχιών και υπάρχει έτσι δυνατότητα για τους πιθανούς αποδέκτες να πάρουν πληροφορίες από αυτά τα σημεία υποστήριξη είναι το πρώτο σημείο επαφή για τον απλό πολίτη. Υπάρχει και μια συμβουλευτική δομή. Οι εταίροι συνεδριάζουν πέντε φορές κάθε χρόνο για να παρακολουθήσουν την εκτέλεση του προγράμματος και επίσης το γραφείο του εκτελεστικού προγράμματος έχει την ίδια χρονική ε, συχνότητα για τις ε, για τις συναντήσεις του. Έχουμε λοιπόν ένα οργανόγραμμα το οποίο είναι λίγο δύσκολο να το διαβάσετε στην οθόνη, μόνο σε χαρτί μάλλον θα μπορείτε να το διαβάσετε. Σας έχω παρουσιάσει βέβαια τα βασικά στοιχεία. Έχουμε μια εποπτική αρχή η οποία ελέγχει τη διαχειριστική αρχή και κάθε πόλη και γενικά η περιφέρεια η δυτική έχει και μια ομάδα η οποία είναι συμβουλευτική είναι ομάδες που περιλαμβάνουν τους εμπλεκόμενους, οι επιχειρήσεις, ε, εμπορικά επιμελητήρια, πανεπιστήμια, σε διάφορα επίπεδα χάραξης πολιτικής. Βλέπετε και πάλι μία άλλη την οργάνωση του συστήματος και ερχόμαστε τώρα στο, στην επόμενη διαφάνεια. Πώς ε, Επέτυχε λοιπόν αυτή η στρατηγική παρά το γεγονός ότι χρειαστήκαμε δύο χρόνια για να την διαπραγματευτούμε και ήταν δύσκολες διαπραγματεύσει, γιατί έπρεπε να δημιουργηθεί ένα κλίμα αμοιβαία εμπιστοσύνη και ανάληψη ευθυνών. Τελικά υπήρξε μια συμφωνία. Τα μνημόνια κατανόηση λοιπόν είχαν συνταχθεί μετά από δύο χρόνια και μπορούσαμε να ξεκινήσουμε χωρίς να υπάρχουν διαμάχες για το ποιο είναι αρμόδιος για ποιο τμήμα της εφαρμογής. Αυτή τη στιγμή περίπου 65% του προπολογισμού βρίσκεται δεσμευμένο για συγκεκριμένα σχέδια. Έχουμε απλώς πρακτικά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε όπως σε όλα τα άλλα προγράμματα. Η απόδοση των σχεδίων ήταν αρκετά καλή και δεν υπήρξαν παράπονα και διαμαρτυρίες σε σχέση με την ποιότητα και την ποσότητα των σχεδίων. Φυσικά όμως πρέπει να συνεχίσουμε να αποδίδουμε την πρέπουσα προσοχή σε όλα αυτά. Χρειαζόμαστε λοιπόν την επίσημη περαιτέρω εκχώρηση, όπως αναφέρει ο κανονισμός. Όταν θέλουμε λοιπόν να βρούμε μια λύση, πάντα πρέπει να στρεφόμαστε στον κανονισμό 1083-2006 και φυσικά ο στόχος μας είναι πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την ε, θέση που αφορά ο κανονισμό, που ε, μάλλον θεσπίζει ο κανονισμός, με μια αποκεντρωμένη λειτουργία στην πράξη, ώστε κάθε πόλη να μπορεί να λύνει τα προβλήματά της. Ο κανονισμός δεν ήταν το μόνο σημείο κίνησης αλλά μας βοήθησε σε μεγάλο βαθμό και ήταν εύκολη η εφαρμογή τους στις τομές της δικές μας και η χρήση τους στο κύριο πρόγραμμα. Το επόμενο τώρα. Χρησιμοποίησαμε και άλλο ένα κανονισμό. Για τον κανονισμό μάλλον για την ε, διατύπωση που αφορά τις συνολικές χορηγήσεις σε σχέση με την προτεραιότητα 3 σε επίπεδο πόλης και εδώ χρησιμοποιήθηκε ο μηχανισμός εκχώρησης. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι η διαχειριστική αρχή είναι αυτή η οποία είναι σε τελική ανάλυση και η υπόλογη. Η αποκεντρωμένη δομή λοιπόν μπορεί να έχει λειτουργήσει σημαντικά σε καθημερινό επίπεδο και βασίζεται σε ε, σωστή κοινή ανάλυση κινδύνων και αμοιβαία ε, συνεργασία, αλλά εξακολουθεί η διαχειριστική αρχή να είναι υπεύθυνη. Εδώ βλέπετε το πώς κατανέμονται τα κονδύλια αναπεριοχές. Αυτός δεν είναι ο νομικά δεσμευτικός προϋπολογισμός, είναι τα επίπεδα χρηματοδότηση τα οποία χρειάζονται για να υπάρξει χρήση χρηματοδότηση από, τα τοπικά, από τους τοπικούς προϋπολογισμούς. Και τέλος, η Κατευθυντήρια Επιτροπή και η Εποπτική Αρχή είναι αυτές που τις ανέφερα προηγουμένως. Επομένως μπορώ να κλείσω αυτή την παρέμβαση και είμαι, είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λαμβάνει υπόψη την ειδική θέση των πόλεων μέσα σε ένα γενικό πρόγραμμα και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε στο μέλλον <clears throat> να χρησιμοποιήσουμε και καλύτερα το μηχανισμό της Τζέσικας και να βρούμε και άλλους τρόπους χρηματοδότησης πέραν των χορηγήσεων που θα μπορούσαν να είναι σημαντικές. Και μπορείτε να φανταστείτε μηχανισμούς που να χρησιμοποιούν μοντέρνα χρηματοοικονομικά εργαλεία όπως η Τζέσικα που είναι πιο χρήσιμα ίσως από τα στοιχεία του προγράμματος Urban στο παρελθόντος. Αυτή τη στιγμή τη χρονική η μεγάλη δυσκολία να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ολοκληρωμένα προγράμματα για τις ε, ε πόλεις. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου και κονδύλια από άλλα ταμεία συγχρόνως και πιστεύω ότι όταν ε, συγκεντρώσει κανείς και συνδυάσει τα χρηματοοικονομικά εργαλεία με εργαλεία όπως το Τζέσικα στο χρηματοοικονομικό τομέα και με τη δυνατότητα εκχώρησης σε ενδιάμεσους φορείς έχουμε πολύ καλές προοπτικές για να εφαρμόσουμε ολοκληρωμένα προγράμματα τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν με ενδιάμεσους φορείς όπως είπα και με εκχώρηση εποφελώς τα κονδύλια αυτά. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Thank you very much. Ευχαριστούμε. Νομίζω θα ήταν καλύτερα εάν τώρα θέταμε τα ερωτήματα, ίσως τρία και έπειτα να περνάγαμε στην επόμενη παρουσίαση. Ο κύριος Φανίστερου, Με συγχωρείτε πρέπει και εγώ να παρέμβω, γιατί έχουμε κατάλογο αγορητών. Συμφωνήσαμε λοιπόν να έχουμε τρία ερωτήματα. Πρώτα, απαντήσεις. Ωραία. Ο κύριος Φαλίστερο, η κυρία Ντέλη και ο κύριος Φαϊμός. Ένα πολύ σύντομα, σύντομο ερώτημα. Γιατί μπορέσετε να διαχειριστείτε την υπεκχώρηση της συγκεκριμένη στις κατοχώρες και αυτό δεν πέτυχε τόσο πολύ στην υπόλοιπη Ευρώπη. Υπήρχε παράδοση ούτως ή άλλως της πόλης της Ολλανδίας να λειτουργούν ως αστικά κέντρα, να καταρτίζουν προγράμματα. Μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα για άλλους. Το συγκεκριμένο Ολλανδικό παράδειγμα για την υπεκχώρηση. Για να αποφύγουμε και μια διετία συζητήσεων, ίσω μπορείτε να μα πείτε το μυστικό σα. Η κυρία Αντέλη. Θα ακούσουμε τα τρία ερωτήματα, έτσι. Νόμιζα ότι θα έχουμε ακούσει τις δύο παρουσιάσεις πριν ε, ερωτήσουμε. Θα κάνω στο τέλος την ερώτησή μου, λοιπόν. Ο κ. δεν είναι εδώ. Όχι είναι. Θέλετε να παρέμβετε τώρα ή μετά. Γιάννη. Έχουμε μόνο την ερώτηση του κυρίου Φανίστελ τελικά. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας ε, δώσω εγώ το μυστικό των κατοχωρών. Πάντως είναι ένας συνδυασμό τριών πραγμάτων που λειτουργήσαν στη χώρα, στη χώρα μα και όχι ίσως σε άλλες που δεν τον ξέρω. Ένα είναι η ιστορική κληρονομιά μας. Υπήρχε πραγματικά πάντοτε ειδικό ρόλος ιδιαίτερος για τις πόλεις και μια περίοδος προγραμματισμού για τα αστικά κέντρα με, συγκεκριμένο, με συγκεκριμένη προσέγγιση για το διάστημα 2000-2006. Ήταν συνηθισμένες λοιπόν οι πόλεις της Ολλανδίας. Επίσης, λόγω του συστήματος των κατεχωρών είναι πολύ επακεντρωμένη η λειτουργία των πόλεων, ιδίως στα δυτικά. Βοήθησε αυτό γιατί μέχρι τώρα είχαν έλλειψη συνεργασία και ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα να υλοποιήσουν τα του προγράμματος. Και επίσης πολύ σημαντικό, κάτι που σα λείπει από άλλε χώρες, είναι όταν υπάρχει υψηλό βαθμό αποκέντρωση, υπάρχουν και πολλά συστήματα, όπω συστήματα τεχνολογιών και πληροφορική και συστήματα τα οποία μπορεί να κατεβάσει κανεί από το διαδίκτυο και πολλοί κανόνες ε, επιλεξιμότητας. Άλλοι για το Άμστερνταμ λόγου χάρη, άλλοι για το Ρότερνταμ. Άρα δεν υπήρχαν σοβαρέ αντιπαραθέσει ή αντιφάσεις που έπρεπε να επιλύσουμε. Δεν χρειάστηκε οκτώ εταίροι να συμφωνήσουν σε ένα πρόγραμμα εθνικό επιλεξιμότητας. Χρησιμοποίησαμε το εθνικό μας ε, το νομοσχέδιο περί επιλεξιμότητας το ε, ενιαίο σύστημα τεχνολογίας για πληροφορικής, δεν προσθέθηκε διοικητικό άχθος και νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει και σε άλλες χώρες. Κάποιοι το φοβούνται πολύ, από ό,τι ακούω, το περαιτέρω διοικητικό άχθος. Με τόσα διαφορετικά διοικητικά συστήματα, τα συστήματα υπολογιστών, εμείς δεν το αντιμετωπίσαμε αυτό. Καταφέραμε να το παρακάμψουμε. Πολύ ωραία. Και τώρα να προσκαλέσω τον κύριο Μούλιγκαν να μα κάνει την παρουσίασή του για να περάσουμε μετά στη γενική συζήτηση. Thank you, Madam um, and thank you for Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρότασή σας, πρόσκλησή σας να παρουσιάσω τα στοιχεία αυτά που έχουν μεγάλη σημασία για την ανάπλαση της πόλης του Belfast και για το πώς λειτουργούν τα Ευρωπαϊκά Διευθυντικά Ταμεία. Στα επόμενα 10 με 15 λεπτά θα προσπαθήσω να δώσω έμφαση σε ένα μέρος από το έργο του Landing και να πω ότι αυτό που θεωρώ ότι συνετέλεσε στην επιτυχία μας, να σας παρουσιάσω δηλαδή ποια ήταν αυτά τα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα να πω ότι το Belfast τον 20ο ε, αιώνα ήταν ε, μια ιδιαίτερα βιομηχανική περιοχή με, με ναυπηγικά ε, εργοτάξια, με με ιδιαίτερα προβλήματα ρήπανση και παρόλα αυτά διαθέτει ένα εργατικό δυναμικό πολλέ φορέ με ιδιαίτερε δεξιότητε, αλλά όχι τόσο προσαρμοσμένο στη σύγχρονη οικονομία και τι ανάγκε τη. Επίση, η πόλη είχε ουσιαστικά στρέψει τι πλάτε τη στον ποταμό Λάγκαν και υπήρχαν προβλήματα κυκλοφοριακού κίνησης και βεβαίως συμφόρησης και ρήπανσης. Οι δεξιότητε τώρα του εργατικού δυναμικού ε, άρχισαν να λείπουν όταν έφευγαν οι άνθρωποι και όταν ε, έτεινε να διωγγώνεται ο δημόσιο τομέα. Και δεν υπήρχε και μεγάλη εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων ε, στην περιοχή. Ίσως με μερικές φωτογραφίες να δείτε πώς είχαν τα πράγματα τότε. Βλέπετε επίσης βλέπετε ότι υπήρξαν επιθέσεις στο εμπορικό κέντρο της πόλης το ίδιο. Και τα προβλήματα δεν ήταν μόνο ανθρωπογενή. Ο ποταμός Λάγκαν είναι ένας ποταμός που έρεε στο πλάι της πόλης και πολλές φορές υπήρχαν προβλήματα και με πλημμύρες από τη λάσπη. επειδή το Belfast εξαρτήθηκε από την ε, επεξεργασία του άνθρακα ε, αέριο για πολλά χρόνια, υπήρχαν προβλήματα ρήπανσης στον ποταμό. Εδώ βλέπετε ότι μερικές εικόνες ε, της πόλης που παρά την υποβάθμιση που υπήρχε, κάποιοι δεν είχαν χάσει την εμπιστοσύνη τους της πόλης να αναβιώσει, να αναγεννηθεί. Αυτή η φωτογραφία έχει πάρθει από το αστικό κέντρο του Belfast και από το σχετικό πρόγραμμα για την αστική περιοχή του Belfast του 1987, όπου υπήρχε ήδη ένα πρόγραμμα ανάπλασης. Η κυβέρνηση ήδη επεξεργάστηκε ένα πρόγραμμα για τον ποταμό Λάγκαν για να δει πώς μπορεί να συμβάλλει η αξιοποίηση του ποταμού στην αναπλάση της πόλης. Και την ε, ευθύνη αυτή ανέλαβε ακριβώς ανεξάρτητος φορέας από το 89 ε, η Ένωση για τον ποταμό Λάγκενσάιτ. Και τα έργα του οργανισμού αυτού ολοκληρώθηκαν το 2007, αλλά από την ίδρυσή του το 89 ο οργανισμός αυτός συνένωσε τις δυνάμεις της κοινότητας ώστε να συνδράμουν ε, τα έργα τους στην περιοχή για την οποία ήταν υπεύθυνοι και να δώσουν τελικά μια νέα ζωή σε αυτή την περιοχή. Υπήρχε συγκεκριμένο στόχος και εντολή να να αναπλαστεί συγκεκριμένη περιοχή προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δημόσιες και ιδιωτικούς επενδυτές να δημιουργήσει ένα ελκυστικό περιβάλλον για κατοίκηση και για ψυχαγωγικού σκοπού. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο λοιπόν πλαίσιο για το Λάγκενσάιντ, για την ευμερία των ε, ανθρώπων, των πολιτών, των επιχειρήσεων και του ίδιου του, της, της ίδιας τοποθεσίας. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε περίπου ποια είναι η περιοχή για την οποία ήταν υπεύθυνο ο οργανισμός για το Λάγκενσάιντ. 150 εκτάρια ήταν αρχικά αυτή η επιφάνεια η οποία επεκτάθηκε μετά την ίδρυση του οργανισμού 10 χρόνια μετά, ώστε να προσθεθούν περίπου 200 εκτάρια ακόμη από την περιοχή της πόλης. Η αρχική προσέγγιση τώρα ήταν τι θα γίνει ακριβώς με την ίδια την ε, υποδομή, τις ίδιες τις υποδομές της περιοχής, προκειμένου οι πολίτες ε, στο περιβάλλον αυτό να μπορούν να κατοικούν, να επενδύουν και να ψυχαγωγούνται. Βεβαίω, το θέμα ήταν πώ θα αντιμετωπίζαμε και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπω τη ρήπανση και των πλημμυρών, και να δημιουργηθούν οι κατάλληλε υποδομέ και για απορρίπανση του ποταμού με την ε, επεξεργασία των ε, λιμάτων, τι εγκαταστάσει ε, φυσικού αερίου και τη δημιουργία δρόμων, πεζοδρόμων και το καθεξής. Εδώ βλέπετε κάποιε από τι ιδέε που αναπτύχθηκαν χάρη και στα διαφορετικά ταμεία με νέα, με σύγχρονα προγράμματα μηχανικής. Εδώ βλέπετε να έχει γίνει πρόβλεψη μέχρι και για τους σολομούς και το πώς θα ανέβουν το ρεύμα του ποταμού για να φτάσουν στους στόχους αναπαραγωγής τους. Όλα αυτά στα πλαίσια ανάπλασης του ποταμού Λάγκαν. Εδώ βλέπετε χέρσωση, μέρος χέρσωσης του ποταμού και η προσέγγιση τώρα που αναπτύχθηκε από το 1995 ήταν να αναγνωρίσουμε ότι έπρεπε να διασυνδεθούν καλύτερα οι ανάγκες της κοινότητας και της εργατικής δύναμης, του εργατικού δυναμικού που κατοικούσε γύρω από την περιοχή του Λάγκαν. Οπότε η στρατηγική μας βασίστηκε στις ανάγκες αυτής της κοινότητας. Αλλά θέλαμε να δώσουμε και νέα ζωή σε αυτή την περιοχή. Και από το 1997 υπήρχε και μια στρατηγική με συγκεκριμένα γεγονότα που λαμβάνονταν υπόψη στο σχεδιασμό μα. Όλε αυτέ οι στατικέ λοιπόν οδήγησαν στο να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή στην εταιρική σχέση και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου και σε επίπεδο αρχών τοπική αυτοδιοίκηση και φορέων των ε, πολιτών. Εδώ έχετε μια ανακεφαλαίωση των επιτευγμάτων μας. Στα περίπου 20 χρόνια, 30 χρόνια λειτουργίας μας, περίπου είχαμε ένα σχεδόν δις ε, επενδύσεων, με αναλογία 1,5 στήριξης από τον ιδιωτικό τομέα. Δημιουργήθηκαν 14.000 θέσεις εργασίας, ε, πολλά, πολλοί χώροι λιανικής πώληση και χώροι ψυχαγωγικοί και επίσης κατοικίες. Βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια πόσο κοντά βρίσκονται ε, οι κατοικίες των πολιτών ε, στην περιοχή του Λάγκερσάιντ. Βλέπετε εδώ ένα θέατρο το οποίο είναι ακριβώς δίπλα στο ποτάμι, αλλά υπάρχει ακριβώς ε, παραπέρα μια γειτονιά με αρκετά μειονεκτούσα, η οποία ονομάζεται Markets και εξηγιάνθηκε και αυτή χάρη σε κονδύλια που αξιοποιήσαμε. Δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως συσχετίστηκε η ανάπλαση του Λάγκενσάιντ με τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας. Κάτι άλλο που ήταν σημαντικό ήταν ότι οικοδομήθηκε και μία γέφυρα στην περιοχή ελιμενισμού και δημιουργήθηκαν και κατάλληλες εγκαταστάσεις από κάθε όχθη και στις δύο όχθες του ποταμού και ο σκοπός εδώ ήταν να απομακρύνουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα από το κέντρο της πόλης. Και τώρα πολύ σύντομα να σα δείξω κάποιες φωτογραφίες που ίσως να σα δώσουν μια εικόνα για την ποιότητα του έργου που επιτελέσαμε. Εδώ βλέπετε κάποια εντυπωσιακά συγκροτήματα κατοικιών δίπλα στο ποτάμι. Ε, δεν είναι όμω μόνο νέα κτίρια που χτίστηκαν, αλλά και κάποια παλιά που αναπαλαιώθηκαν. Και αξιοποιούμε εδώ και την περιοχή των ε, προβλητών της όχθης του ποταμού. Την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που είχε. Και στις επόμενες διαφάνειες πολύ γρήγορα βλέπετε εικόνες από το, τη σημερινή μορφή της περιοχής. Τώρα, τι θεωρούμε ότι ήταν αυτό που συντέλεσε στην επιτυχία μας. Ποιοι ήταν αυτοί οι παράγοντες που μας επέτρεψαν να πετύχουμε είναι ευρέως αποδεκτή η επιτυχία του πειράματό μας και από έρευνα του ΩΣΑ πρόσφατα εντοπίζεται αυτό με πολύ θετική αποτίμηση του έργου του οργανισμού του Σάιτ. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπήρχε ένα κυρίαρχο πρόγραμμα, ένα βασικό πρόγραμμα στο οποίο βασιστήκαμε. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν πολιτικοί ηθήνοντες, αξιοποιήθηκε η συμβολή από ε, λειτουργούς της τοπικής αυτοδιοίκηση μέχρι υπουργού που συμμετείχαν στην επιτυχία μας. Επίσης υπήρχε πολύ συγκεκριμένη, στοχευμένη εντολή Μπορώ να το διαβεβαιώσω εγώ για την περιοχή του Λάγκενσάιντ, την οποία εργάστηκα εγώ ίδιο. Υπήρξαν επίση δυνατότητε εξαγορά γη και ένα, πολύ, ένα τοπικό συμβούλιο με πολύ μεγάλη επιρροή. Επίσης, η σταδιακή εξυγένση των υποδομών και η σταδιακή μας που βασίστηκε στις ανάγκες της τοπικής κοινότητας με τη συνδρομή των διευθυντικών ταμείων και του Κοινωνικού Ταμείου και των Ταμείων Περιφερειακής Ανάπτυξης, όλα αυτά συνετέλησαν στην επιτυχία μας. Τώρα κάποιες τελευταίες φωτογραφίες. Δείτε την ε, διαφορά. Πρώτη φωτογραφία, ο ποταμός όπως ήταν πριν, τώρα οι πλημμύρες που σας είχα δείξει στην αρχή. Ξαναδείτε την πρώτη, πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο. Και άλλη μια σύγκριση του πριν και του μετά. Η παρακμή που σας ανέφερα προηγουμένως, η υποβάθμιση πριν την ανάπλαση. Δείτε τώρα πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα με την επόμενη φωτογραφία. Σε αυτό το μπαρ να μην παραλείψετε να πάτε να έρθετε στον Belfast. Να ολοκληρώνοντας λοιπόν να πω ότι η κληρονομιά που μας αφήνει το Lagenfeld από το 2007 δεν μπορεί να ε, υποτιμηθεί. Ε, δημιουργήθηκε ένα φυσικό εργασιακό περιβάλλον όπου το εθνικό και ξενοκεφάλαιο ήταν πρόθυμο να επενδύσει και μάλιστα σε μια από τις πιο ταραχώδες περιόδους της ιστορίας μας. Αλλά ενώ ήταν ένα κίνητρο για την γενικότερη αναβίωση και ανανέωση της πόλης, το Λάγκενσεντ αποτελεί παράδειγμα για τη Βόρεια Ιρλανδία και τον Μπέλφαστ γενικότερα. Δηλαδή δείχνει πώ μπορούμε να πετύχουμε ένα πιο πολιτισμένο, πιο ε, πρόσφορο μέλλον με τι κατάλληλε προσπάθειε. Υπάρχουν όμω ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν στον Μπέλφαστ, όπω με την ανεργία, με την οικονομική ανάπτυξη που έχει τελματωθεί, ε, με τι επενδύσει. Το Lagenside ήταν ένα πρόγραμμα που εάν ε, μας οδηγήσει σε μίμηση με άλλα παραδείγματα μπορεί να βοηθήσει την εξέλιξη πολλών πόλεων και στην Ευρώπη και αλλού. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μισή ώρα για τη συζήτηση και θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ, Ο επικεφαλής μονάδας για την αστική ανάπτυξη και εδαφική συνοχή και ο Σαντιάγο Ρίβας που είναι υποδιευθυντής του τμήματο αυτού Λοιπόν, όποιος θέλει να πάρει το λόγο είναι ευπρόσδεκτος. Πρώτα απ' όλα, Καρίμα Ντέλη. Η πρώτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Βλάσα, σα ευχαριστώ για αυτή την ε, πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση. Αυτό που απορρέει από όλα αυτά είναι ότι για να αποφευθεί ο κίνδυνος κατακαιρματισμού της πολιτικής συνοχής και να είναι ολοκληρωμένες οι πολιτικές για την κοινωνική συνοχή, χρειάζεται να βασιστούμε στις πόλεις σήμερα που θα είναι πραγματικοί φορείς που μπορούν να εφαρμόσουν αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις μεταφορές, για την ενέργεια, για το κλίμα, την καταπολέμηση της φτώχεια κλπ. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εκείνη που ε, είναι στην πρώτη γραμμή για την εφαρμογή των μέτρων. Βλέπουμε από αυτά τα προγράμματα ότι μπορεί να εφαρμοστούν συγκεκριμένα μέτρα για την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η πολιτική της συνοχής λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι μια πολιτική με τις πόλεις και όχι για τις πόλεις. Θα πρέπει αυτό να ε, ληφθεί υπόψη και να ενταχθεί σαν ιδέα. Λοιπόν, για να σας βοηθήσουμε κύριε Βλάσα για την πολιτική σας έκθεση, λέει και ότι θα πρέπει να ρίξουμε μία ματιά και στις νέες προκλήσεις εκεί που θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες οι πόλεις. Πρέπει να καταπολεμήσουν, έχουμε την πρόκληση της αλλαγής του κλίματος. Τα βασικά διακυβευόμενα για την βιώσιμη πόλη είναι να διαπιστώσουν ποιος είναι ο ρόλος τους. Και η μάχη για το κλίμα θα γίνει στις πόλεις, με τις πόλεις. Όπως είπατε, ο μισός πληθυσμό, τα τρία τέταρτα του πληθυσμού, του ευρωπαϊκού πληθυσμού, ζει στις πόλεις, τα τρία τέταρτα εκπομπών διοξιδίου του άνθρακο που έρχονται τι πόλει και 80% της κατανάλωσης ενέργειας ε, γίνεται στις πόλεις. Άρα θα πρέπει να το πούμε και το επαναλαμβάνω ότι η μάχη του κλίματος θα γίνει στις πόλεις. Το βασικό ερώτημα είναι η θέση της διακυβέρνησης θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Εκεί είχαμε διάφορα μέσα στη θέση μας. Ας πάρουμε παραδείγματος χάρη το πρόγραμμα Urban. Βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι λίγο πολύ θετικά διότι καταφέραμε να τονίσουμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ όλων των τοπικών φορέων που, που ακολούθησαν τα προγράμματα. Και αυτό το ζήτησε και η Σύμβαση των Δημάρχων. Είναι σημαντικό λοιπόν πραγματικά να μπορούν να συμβάλλουν όλοι οι φορείς στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Διάβαζα το έγγραφό σας που λάβαμε όσον αφορά τους δίκτες Πρέπει να προσέξουμε συνάδελφοι. Εγώ είμαι από μια πόλη, Ile de France, μια περιοχή της Γαλλίας στο Παρίσι, η Ile de France έχει υψηλό ΑΕΠ και υπάρχουν πάρα πολλές κοινωνικές διαφορές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στην πολιτική συνοχή. Και θα ήθελα να πω ότι βλέπουμε να γίνουν επενδύσεις όσον αφορά τεχνική αρρωγή υπενθυμίσατε πριν ισχύσουμε το Τζέσικα και την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κλπ. Πράγματι, αλλά θα πρέπει να δοθούν οι πόροι κατάλληλοι. Και όσον αφορά την ενέργεια, πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Σας δίνω μια ιδέα. Αστική ενέργεια Εκεί πρέπει να κινηθούμε, να δούμε πώς γίνεται η διαχείριση ενέργειας στην πόλη. Είδαμε το ΦΕΝΤΕ δίνει 4% για τα κτίρια στην Ευρώπη. 21% από τους πόρους αυτούς χρησιμοποιούνται. Θα ήθελα να ξέρω ποια εργαλεία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τελικά, ούτως ώστε όλες οι χώρες χρησιμοποιούν τα χρήματα για την ενεργειακή απόδοση, κυρίως τα κτίρια, και να καταπολεμήσουμε την, ε, τον, ε, τον ανασφαλή εφοδιασμό τον ενεργειακό. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα νέα εργαλεία, τα σωστά εργαλεία. Αν χρησιμοποιήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία, νομίζω ότι θα πετύχουμε το στόχο και νομίζω ότι θα σας υποστηρίξουμε στην πολύ καλή σας έκθεση κύριε Μπλάζα. Και έχουμε 7 συναδέλφους στον κατάλογο. Παρακαλώ να είστε όσο σύντομοι γίνεται. Ο Πίτερ Σάιμον είναι ο επόμενος που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο από την Ολλανδία, ιδίω γιατί στη Γερμανία δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει τέτοια κατανομή αρμοδιοτήτων στα ομοσπονδιακά κρατήρια που δεν μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια οδό. Πολλές φορές αναγκάζονται λόγω της δομής αυτής τα ομοσπονδιακά κρατήρια να ακολουθούν οδούς που δεν ανταποκρίνονται πάντα στο συμφέρον του πληθυσμού. Αν ήταν ενδιαφέρον το θέμα αυτό της ε, περαιτέρω ε, εκχώρησης. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν νέους χώρους για συνεργασία, για δράση της αγοράς, να υπάρξει συνέργεια μεταξύ ε, οικονομικών και βιομηχανικών φορέων όταν θέλουμε να προωθήσουμε την ανανέωση των πόλεων. Αλλά κύριε Φλάσεκ, θέσατε σωστά το ερώτημα πού βρίσκεται το όριο. Μέχρι πού πρέπει μια πόλη να αναλάβει την ε, εφαρμογή προγραμμάτων που έχουν τέτοιο χαρακτήρα. Όταν έχουμε μια πόλη η οποία έχει παραγωγή 20.000 πολίτες μονάχα και 6 εκατομμύρια χρηματοδότηση από το Urban, βρισκόμαστε στα όρια της δυνατότητας να λειτουργήσουν τέτοια προγράμματα. Επίσης, πρέπει να δούμε ποιο είναι το μέγεθος το οποίο επιτρέπει να υπάρχει αυτός ο λειτουργικός χώρος. Επίσης, να λάβουμε υπόψη τη δυνατότητα η εκ, νέο εκχώρηση να γίνεται και σε ευρύτερου φορεί, όπως στην περίπτωση της Ολλανδίας που αφορούσε μεγάλες πόλεις. Επίσης, για τα θέματα της εταιρικής σχέσης που αναφέρθηκαν από εσά. Είναι απαραίτητο να δούμε ότι και εδώ, και εγώ γνωρίζω καλύτερα τη δική μου χώρα, χρειάζεται μια εταιρική σχέση για να υπάρξει η ανάπτυξη των λειτουργικών προγραμμάτων. Στη Γερμανία όμως αυτό δεν έχει γίνει πραγματικότητα. Ούτε στη σύλληψη των προγραμμάτων, ούτε στην εκτέλεσή τους. Γι' αυτό δεν λειτουργεί και η συγχρηματοδότηση. Γιατί δεν υπάρχει συνοχή που να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση ακριβώς αυτών των ενεργειών που είναι οι σημαντικές για το τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό τονίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχει ο τοπικός παράγων χωρίς αυτό να κάνει πιο δύσκολη, πιο πολυδέδαλη και πιο άκαμπτη τη διαδικασία. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε μια σειρά από κριτήρια τα οποία θα αντιμετωπίσουν την ανάγκη να καθορίσουμε πώς θα συμπλέκονται τα διάφορα επίπεδα και με ποιο τρόπο μπορεί να συμμετέχει το τοπικό επίπεδο στην εκπόνηση και την εφαρμογή των ε, προγραμμάτων. Αλλά αυτός ο κατάλογος πρέπει να επιτρέπει και μία διεύρυνση. Στη Γερμανία έχουμε τη δομή αυτή από την, ε, έχουμε την κυβέρνηση και τα ομοσπονδιακά κρατήρια. Τα ομοσπονδιακά κρατήρια όμως θα πρέπει να έχουν κριτήρια εκχώρησης σε υποκείμενους φορείς όπως είναι οι πόλεις και οι επαρχίες. Χωρίς αυτό να οδηγήσει σε ένα πρόσθετο γραφειοκρατικό άχθο για, ε, για τα προγράμματα αυτά. Και το τελευταίο σημείο που αναφέρατε, την ολοκληρωμένη σχεδίαση. Νομίζω ότι τα ερωτήματα που θέλετε, θέτετε είναι ακριβώς τα σημαντικά γιατί αυτά είναι ερωτήματα που με ταλανίζουν και εμένα. Θέτετε λοιπόν το θέμα για το ποιοι πρέπει να είναι οι κανόνες του παιχνιδιού για την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων και σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να λειτουργήσει η ολοκληρωμένη σχεδίαση από τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, στη Γερμανία μπορώ να σας πω και πάλι, τα πράγματα δεν είναι απλά. Εάν θέλουμε ολοκληρωμένη δράση θα πρέπει να υπάρχουν πιο δεσμευτικοί κανόνες και θα πρέπει να είναι και σαφείς και να μπορούν να λειτουργούν με ακρίβεια. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη κύριε Τσίμερ που έκανα αγγλοσαξονικό το όνομά σας. Ο Γιάνν Όλμπριχτ έχει τώρα το λόγο. Ναι. Ένα πάρα πολύ σύντομο ερώτημα και στους δύο μιλητές. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν τις νέες λύσεις και έχουμε και τις εμπειρίες του παρελθόντος. Ενώ συζητάμε αυτή την ε, ανάθεση των ε, καθηκόντων, την εκχώρηση καθηκόντων, τα λειτουργικά προγράμματα είναι καλύτερα για τις πόλεις, για μια πόλη ή για μια ομάδα πόλεων ή καλύτερα να έχουμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την περιφέρεια ή για μεγαλύτερη έκταση με εκχώρηση στις πόλεις. Τι είναι καλύτερο, να επιφορτίζεται η πόλη με το λειτουργικό πρόγραμμα ή να γίνεται υπό εκχώρηση αν θέλετε. Ανδρέα ε, Πάνω απ' όλα θα ήθελα να εκτιμήσω και τις δύο παρουσιάσεις που έγιναν εδώ ε, και μας έδωσε συγγητής μια εικόνα για το πρόγραμμα το ευρωπαϊκό για τα αστικά θέματα. Θεωρώ αυτή τη συζήτησή μας θεμελιώδου σημασίας για την ανάπτυξη της πολιτικής συνοχής. Πιστεύω ότι η πολιτική συνοχή στα επόμενα χρόνια, μάλιστα όταν θα συζητήσουμε και στα πλαίσια των δημοσιονομικών προοπτικών το θέμα, θα απαιτήσει πάρα πολύ ένα μεγάλο στοιχείο καινοτομίας πολύ καινοτομία. Και αυτή η καινοτομία περνά από την πρόκληση την αστική. Είναι η βασική πρόκληση που έχει μπροστά τη η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Την πρόκληση των πόλων. Αν θέλουμε να είναι και αξιόπιστη στόχη που έχουμε θέσει, φέτο με την πολιτική του 2020, αυτή η πολιτική ε, βρίσκει την εφαρμογή της και την υλοποίησή της στις πόλεις μας, στις πόλεις της Ευρώπης όπου εκεί συγκεντρώνεται το 80-85% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και έχουμε 70-75% παραγωγής ΑΕΠ. Ε, πιστεύω λοιπόν πραγματικά μία από τις βασικές προκλήσεις των επόμενων ετών που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Και το, το σχέδιο εκθέσεως και οι παρουσιάσεις που έγιναν και οι παρουσιάσεις εμπειριών είναι αρκετά σημαντικά θέματα και θα ήθελα να συνεργαστώ τα μάλα και εγώ για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε κοινέ προσπάθειε σε επόμενε εβδομάδε, σε επόμενου μήνε. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε άλλα δύο μεγάλα θεμελιώδη ζητήματα. Από τη μία πλευρά κάτι που ήδη υπόθηκε. Από πλευρά νομική, πώ τροποποιούμε του κανονισμού. Διότι αυτή είναι βασική η προπόθεση. Αν θέλουμε να δώσουμε αξιοπιστία σε αυτέ τι ε, πολιτικέ. Παραδείγματο χάρη, θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό ε, τη γενική γενικής που, αφορούσε τις τρεις πόλεις που ενώθηκαν. Αυτό είναι αξιόπιστο, εφικτό και σε άλλα σχήματα. Θα μπορούσε αυτό το πείραμα υλοποιηθεί και αλλού. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε με προσοχή. Γιατί αλλού εφαρμόζεται σε σημείο αναφορά στο περιφερειακό σύστημα όσον αφορά τη διαχείριση και τη διακυβέρνηση αυτών των μορφωμάτων. Τρίτον, Άλλο μεγάλο θέμα που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι όταν εφαρμόζουμε τα προγράμματα αστικής αναγέννησης ε, και ε, αλλαγή τμήματων μεγάλων των πόλων δεν αρκούν ούτε οι εθνικοί πόροι ούτε οι ευρωπαϊκοί δημόσιοι πόροι. Χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε και να προσελκύσουμε ιδιωτικούς πόρους. Όμως αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Διότι υπάρχει ένας κίνδυνος γνωστός που γνωρίσαμε αυτά τα χρόνια νέων μορφών χρηματοπιστωτικής κερδοσκοπίας ε, που μπορούν να παρισφρήσουν σε αυτά τα προγράμματα αναγέννησης των πόλων. Άρα είναι θεμελιώδη σημασία και από αυτή την έποψη εμείς να βρούμε μορφές υλοποίησης διαφανής, διότι, διότι θέλουμε συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον αφορά τους πόρους για να εφαρμόσουμε πολιτικές αναγέννησης των πόλεων της εμβελίας που συζητούμε σήμερα εδώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι σημαντική η συζήτηση που ξεκίνησε ο εισηγητή και που ξεκινά επίσης και από τι παρουσιάσει που έγιναν. Όλοι πιστεύω ότι είμαστε διαθέσιμοι για να συμβάλλουμε στην διεξαγωγή αυτών των ε, συζητήσεων. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, Ιωσήφ Ματούλα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα πολύ σύντομο Λαμβάνοντα υπόψη ότι έχουμε περιορισμένο χρονικό διάστημα στη διάθεσή μα, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο που άκουσα τι ε, παρουσιάσει αυτέ. Είναι ξεκάθαρο ότι στο επίκεντρο τη πολιτική ε, συνοχή σορεύεται το κεφάλαιο στι μεγάλε πόλει. Μεσαίε πόλει και μεγάλε πόλει. Εκεί βρίσκουμε τον κινητήρα τη οικονομική ανάπτυξη, σε αυτά τα μεγέθη. Το ερώτημά μου είναι, ποια είναι η άποψη όσον αφορά το ρόλο των μικρών πόλεων ή των πολύ μικρών ε, πόλεων για το μέλλον της πολιτικής ε, συνοχής. Για να μην μεγαλώνουμε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ μεγάλων και μικρών πόλεων. Look at the clock, Ρίξτε με και το πόλο. Α, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα μονάχα θέμα. Το πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε όλα αυτά τα σχέδια τα οποία λαμβάνουν χώρα και υλοποιούνται στις διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Κύριε Βλάσακ, αυτό είναι κεφαλαιόδες νομίζω. Όλα τα προγράμματα τα οποία είναι ενοποιητικά, πολιτιστικά και κοινωνικά πρέπει να λάβουν υπόψη όλο τον πληθυσμό. Να λάβουν υπόψη και το δημογραφικό και τον πληθυσμιακό και τον ανθρώπινο παράγοντα. Ένα λεπτό για να μιλήσω και εγώ, λέει η κυρία Χιούμπνερ, θα είμαι η τελευταία ομιλήτρια και μετά ίσως μπορεί η Κομισιόν και οι δύο εμπειρογνώμονε και ο κύριο Φλάσικ να λάβουν το λόγο. όλου. Του έχω αναφέρει όλου. Αυτό που ακούσαμε από τους καλεσμένους μας ήταν κάτι που ονομάζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλή πρακτική. Ο Λαμπέρ Φανίστελ Ρόι ρώτησε σε ποιο βαθμό μπορούν αυτά να μεταλαμπαδευτούν στην Ευρώπη ως βέλτιστες πρακτικές, ιδίως σε δύο τομείς. Ξέρουμε όλοι ότι ανεξάρτητα τα χρήματα που έχουμε στον προϋπολογισμό, εθνικό ή ευρωπαϊκό, δεν είναι ποτέ αρκετά τα δημόσια χρήματα για την αστική ανανέωση και να μπορέσει να αναπτυχθεί ο τομέας, ο αστικός. Οπότε αναφέρθηκε το θέμα των ε, κονδυλίων τα οποία ανανεώνονται, χρηματοδότηση δηλαδή με δάνεια που ανανεώνεται και η Τζέσικα, όλα αυτά που ήταν τόσο χρήσιμα στην ε, Βόρεια Ελλανδία για να ε, προσελκύσουν και ιδιωτικό κεφάλαιο. Ποια είναι λοιπόν τα μέτρα με τα οποία θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε κεφάλαια για την αστική ανανέωση και πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα ποσά λαμβάνοντας υπόψη και τον παράγοντα μόχλευσης που έχουν αυτά τα χρήματα τα οποία προσελκύουν άλλα κεφάλαια. Δεν ξέρω τώρα, ίσως καλύτερα πρώτα τους καλεσμένους μας να, λόγο, να λάβουν το λόγο, μετά η Κομισιόν και μετά ο εισηγητής. Δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε κάποια σχόλια για αυτά που ακούσατε. Είχα ένα συγκεκριμένο ερώτημα που τέθηκε από τον κύριο Όλμπρατ και αναφερόταν σε μένα ρώτησε αν υπάρχει μια δομή η οποία είναι πάντα η καλύτερη, είτε αυτή του προγράμματος City, είτε αυτό της εκχώρησης και επανεκχώρησης. Είναι δύσκολο αυτό να το απαντήσει κανείς για το μέλλον. Θα είναι διαφορετικές οι προκλήσεις, είναι διαφορετικές από αυτές που είχαμε στην πρώτη γενιά προγραμμάτων Urban όπου μας ενδιαφέραν περισσότερο τα κοινωνικά, οικονομικά, ακόμα και τα προγράμματα χωροταξίας ορισμένων περιοχών που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε με την ανάπτυξη. Για το μέλλον τώρα τα θέματα είναι το να μπορέσει να ενσωματωθεί και η πτυχή της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής και όχι μονάχα η οικονομική ανάπτυξη η οποία προκύπτει κυρίως από τις πόλεις. Από αυτή την οπτική γωνία θα είναι πάντα απαραίτητο σαν προϋπόθεση να υπάρχει κάποια επιπλέον εκχώρηση προς τις πόλεις, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο πραγματικά συμμετέχουν στην επίλυση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων, αν θα γίνει σε ένα πρόγραμμα mainstream ή σε ένα ειδικό πρόγραμμα urban. Εγώ θα πίστευα ότι στο κύριο πρόγραμμα, το mainstream πρόγραμμα, θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο και να εξασφαλίσουμε μια διακυβέρνηση σε πολλά επίπεδα, ώστε κάθε επίπεδο να μπορεί να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αυτές και στη συγκεκριμένη περίπτωση η κλιματική αλλαγή και οι ενεργειακές ανάγκες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο σε επίπεδο πόλεων, γι' αυτό πρέπει να είναι στο, στον κορμό του προγράμματος, στο mainstream. Ο συνάδελφός μου όμως ίσως διαφωνεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για να απαντήσω σε ένα ερωτήματα που τέθηκαν για το αν θεωρούμε ότι τα λειτουργικά προγράμματα πρέπει να επικεντρώνονται σε πόλεις ή σε ομάδες πόλεων. Επαναλάβω κάτι που είπα. Οποιαδήποτε προτίμηση για οποιαδήποτε διευθέτηση των διευθετικών ταμείων θα είναι επιλογή των εθνικών κυβερνήσεων. Άρα θα πηχεί κάτι σαν πολιτική στάση και δήλωση. Εμείς απλώς μπορούμε να επισημάνουμε βάσει της ίδιας μας εμπειρίας ότι τα διευθυντικά ταμεία όπως τα διαπραγματευτήκαμε στο πλαίσιο του Λάγκενσάιντ ήταν τόσο ευέλικτα ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα προβλήματα αστικά. Ε, προσαρμόστηκαν δηλαδή στις ανάγκες μας και κάποια από τα μεγαλύτερα προγράμματά μας για τις μεταφορές, ε, το περιβάλλον βασίστηκαν και στις δομές της πόλης. Το να ορίσει κανείς μια περιοχή συγκεκριμένη ως περιοχή του λειτουργικού προγράμματος μπορεί να τα περιορίσει, να περιορίσει τη δυνατότητα ενεργειών σας ε, σημαντικά, όπως σε μια, σε μια μικρή, περιοχή όπως στη Βόρεια Ιρλανδία. Ευχαριστούμε. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ακούσαμε προσεκτικότατα τις παρουσιάσεις και τις ερωτήσεις του κυρίου Μπλάζακ. Θα παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί γνωρίζετε ο Επίτροπος Χάν, όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Λεβαντόφσκι, θα ήθελε να προσέξει όλος ιδιαίτερος τα αστικά ζητήματα είναι από τη Βιέννη και θέλει να τονίσει και εκείνο την αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής. Εκ των υστέρων ε, αξιολόγηση της πολιτικής για, την, ε, για τις πόλεις έδειξε ότι είναι υποφελής ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αστική ανάπτυξη και αυτή η εμπειρία της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης είναι κάτι που αναγνωρίστηκε και ήταν κατευθυντήρια γραμμή της χάρτας της λειψίας που ιδιωθήθηκε από όλους τους υπουργούς για την αστική ανάπτυξη και υποστηρίχθηκε και στη δήλωση Τολέδο. Ήρθε η ώρα που έχει τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Αβώνας που ζητά να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο οι τοπικοί φορείς και οι πόλεις στην αστική ανάπτυξη. Το παίρνουμε αυτό στα σοβαρά και βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των πόλεων. για τα μελλοντικά λειτουργικά προγράμματα. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός με τις περιφέρειες ή με τις εθνικές αρχές. Απλώς πρόκειται περί εκμεταλλεύσεως του δυναμικού κάθε περιοχή στα πλαίσια της εδαφικής συνοχής. Διότι η δαφική συνοχή είναι από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να μην εκμεταλλευτούμε το δυναμικό κάθε περιφέρειας. Και με την πρωτοβουλία για την αστική διάσταση βλέπουμε πόσο κεφάλαιο υπάρχει. Ζητήθηκε άποψη διαφόρων ανθρώπων στην εκ των υστέρων αξιολόγηση. Δεν ήταν τα χρήματα το πιο σημαντικό, είπαν, όσον αφορά την πρωτοβουλία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το πρόγραμμα με τη συμμετοχή των διαφόρων εταίρων. Η Ευρώπη του 2020 βασίζεται σε ολοκληρωμένη ανάπτυξη, με ένταξη. Δηλαδή, οι πολίτες να συμμετέχουν σε κάθε επίπεδο. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση με τη συμμετοχή των πόλων είναι ο καλύτερος τρόπος για την ε, υλοποίηση αυτού του στόχου για την Ευρώπη του 2020. Δεν είναι κάτι που δεν προτείνουμε την υποστήριξη αστική ανάπτυξη μόνο και μόνο γιατί περισσότεροι άνθρωποι ζουν εκεί. Αλλά διότι δημιουργείται έτσι η δυνατότητα η Ευρώπη να μπορέσει να προχωρήσει πιο γρήγορα και να αντιμετωπίσει τις ε, προκλήσεις. Οι πόλεις μπορούν να βοηθήσουν. Ερώτηση τέθη για το ρόλο των μικρών και μεσαίων, μεσαίου μεγέθου πόλεων. Για μας είναι ξεκάθαρο ότι με την εδαφική συνοχή Ζητούμε να ακολουθηθεί η λειτουργική προσέγγιση σε αυτά τα προγράμματα, εφαρμοστούν οι σωστέ στρατηγικέ. Έχουμε δίκτυο μικρομεσαίων πόλεων για την εδαφική συνοχή και θα πρέπει να ετοιμάσουμε στρατηγική για μεγαλύτερες περιοχές και πόλεις. Κυρία Πρόεδρε, ρωτήσατε ποιος ο ρόλος της Τζέσικα και των διαφόρων οικονομικών μέσων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σκέφτεται τώρα σκέφτεται πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το τα διάφορα μέσα εκτός των χορηγιών για τη μελλοντική στρατηγική. Μετά από μια μεγάλη αρχική φάση βλέπουμε επιτάχυνση όσον αφορά την χρήση της Τζέσικα. 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ ε, ήδη έχουν προσημειωθεί και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε φτάσει στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα Θέλουμε να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο το μέσο. Έχετε εγκρίνει τροποποίηση του κανονισμού που αυξάνεται έτσι δυνατότητα χρήσεως αυτών των οικονομικών μέσων για εξοικονόμηση ενέργειας και συναφών μέτρων. Προσβλέπω στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μελλοντικέ προσπάθειες για την διαμόρφωση της πολιτικής συνοχής και θέλουμε οι αστικές περιοχές να παίξουν το ρόλο που τους αρμόζει αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θέλω να απαντήσω σε μέρα από τα σχόλια που ακούσαμε όλοι. Καταρχήν να ευχαριστήσω αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν στην συζήτηση και τον προβληματισμό που έλαβε χώρα, αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ορισμένα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε στη συνέχεια. Μιλήσαμε για την Τζέσικα ως εργαλείο χρηματοδότησης. Πρέπει όμως να κάνουμε και μία σύγκριση για το ποσοστό των χρημάτων που μπορούν να επενδυθούν από τις πόλεις μέσω του μέσου Τζέσικα ώστε να ξέρουν και να μπορούν να προετοιμάσουν και να χρηματοδοτήσουν τα σχέδιά τους. Εμείς στην Τσεχική Δημοκρατία προβήκαμε σε μία ανάλυση που περιέλαβε 620 πόλεις, μεγάλες πόλεις και μικρές πόλεις. Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης είναι 5 με 10% του προϋπολογισμού των πόλεων αυτών μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσα από την Τσέσικα. Και είδαμε τέτοια σχέδια, σαν παράδειγμα, αυτό το οποίο είναι κεφαλαιόδηση είναι να μπορέσει να συμμετάσχει ο ιδιωτικό τομέα και να υπάρξει θέση από κοινού των ιδιωτικών και δημοσίων πόρων. Νομίζω ότι στο μέλλον αυτή θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική και αξιόλογη πηγή χρημάτων και θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Κάτι ακόμα που θέλω να υπογραμμίσω είναι ο ρόλος των εθνικών ενώσεων που των ε, τοπικών αρχών που προβαίνουν σε διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις. Ένα πρόσφορο παράδειγμα είναι οι κάτω χώρες, η Ολλανδία. Αλλά οι πόλεις και οι περιφέρειες μεμονωμένα δεν μπορούν να εξασφαλίσουν καλές συνθήκες, γι' αυτό θα πρέπει να συνενώσουν τις προσπάθειές τους για να έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη και να μπορούν να ασκήσουν από κοινού πίεση στις κυβερνήσεις. Κάτι ακόμα για τους ομιλητές μας για τους βουλευτές δηλαδή που έλαβαν το λόγο, η κυρία Ντέλη αναφέρθηκε στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως ε, η χωμόλυνση, η παρουσία σκόνης, η απουσία πρασίνων χώρων στις πόλεις, οι οχλήσεις από τη μεταφορά κτλ. Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν επίπτωση και στους κατοίκους αλλά και στην ενεργειακή απόδοση και την ε, μείωση της εκπομπής ρήπων. Και φυσικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις κοινωνικές ανισότητες οι οποίες υπάρχουν στις πόλεις. Επίσης, για τις ενεργειακές πηγές δεν μας ενδιαφέρει μονάχα η θέρμανση, αλλά και η ηλεκτροδότηση κτλ. Ναι, λέω στην ε, εκχώρηση και επανεκχώρηση, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε μέχρι ποιο σημείο. Ποιο είναι το σημείο στο οποίο δεν είναι πια πρόσφορο και δεν είναι αποδοτικό το να εκχωρούμε αρμοδιότητες. Και δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε εμεί κάποιο συγκεκριμένο και αυστηρό όριο. Γιατί μπορεί να υπάρχουν μικρές πόλεις οι οποίες έχουν εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα είναι σε θέση να προετοιμάσουν και να εκτελέσουν σωστά σχέδια χρησιμοποιώντας επωφελώς τα κονδύλια. Αλλά για μένα χρειάζεται μια τάξη μεγέθους 100.000 κατοίκων περίπου για μια πόλη να μπορεί να τύχει επωφελούς ε, εκχώρησης. Για τους εταίρους και για την βιωσιμότητα και για την ενδεχόμενη κερδοφορία σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Αυτά πρέπει να είναι σαφή κριτήρια αυτό σημαίνει ότι κάθε σχέδιο θα πρέπει να είναι βιώσιμο στα επίπεδα αυτά και να πρέπει να δίδει και κάποιο κέρδος στους επενδυτές. Επομένως πρέπει να καταδείξει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει αποδοτικά τα χρήματα. Ορισμένοι ομιλητέ αναφέρθηκαν στα χρήματα του ιδιωτικού τομέα. Βεβαίως πρέπει να εμπλέκεται και ο ιδιωτικό τομέα. Ο κύριος Ματτούλα αναφέρθηκε στις μικρές πόλεις. Δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε. Φοβάμαι απλώς ότι πρέπει να σκεφτούμε και περισσότερο για προβλήματα όπως ο πληθυσμός των μικρών πόλεων, ο οποίος μετακινείται για να εργαστεί στις μεγάλες πόλεις και επιστρέφει το βράδυ, οι φοιτητές οι οποίοι πρέπει να πάνε σε μια πιο μεγάλη πόλη να, σπουδάσουν, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι μαγνήτες οι μεγάλες πόλεις, οι οποίες προσελκύουν τους ε, πληθυσμούς, τους κατοίκους από τις μικρότερες πόλεις που βρίσκονται γύρω τους. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών. Και εδώ θα πρέπει να προχωρήσουμε σε συζήτηση και με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό, σε δημοτικό επίπεδο. Ναι, Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τύχουν διαπραγμάτευση στο τοπικό, στο πιο κοντινό προς το πολιτή επίπεδο. Τέλος για το θέμα της μόχλευσης που αναφέρε και η κυρία Χιούμπνερ. Μίλησε για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Τζέσικα προς το σκοπό αυτό. Πιστεύω ότι στο μέλλον αυτά τα εργαλεία θα τύχουν όλο και περισσότερες χρησιμοποίησεις. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να διευκρινίσουμε τις αρχές που διέπουν αυτά τα εργαλεία. Εμείς έχουμε κάνει τις αναλύσεις για τα θέματα αυτά και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι μικρότερες πόλεις και κομοπόλεις δεν έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για το πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί η Τζέσικα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση και καλύτερο επίπεδο γνώσεων μεταξύ αυτών και Εν κατακλείδη, εγώ αναμένω τα σχόλιά σας, γραπτώση με email και εγώ προετοιμάζω το τελικό έγγραφο εργασία. Um, uh, uh, ευχαριστώ πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων για όσον αφορά την έκθεση και ευχαριστώ και τους δύο συναδέλφους από την Ολλανδία και από τη Βόρεια Ιρλανδία, τον κύριο Βαν Ρακ και τον κύριο Ρόμπινσον και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ μπορώ να τη συνεδρίαση και συναντώμεθα με τους αύριο το πρωί με τις κάρτες ψηφοφορίας το πρωί. Παρακαλώ να φύγει το δυνατόν από την αίθουσα διότι έχουμε συνεδρίαση των ε, συντονιστών. Και περιορισμένο χρόνο ως συνήθως ευχαριστώ πολύ εκ νέου και οι συντονιστές σας παραμείνουν στην αίθουσα παρακαλώ.